Ladies uh, και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 3 και 8. Αρχίζουμε δύο λεπτά νωρίτερα δηλαδή, αλλά ας ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση. Σημαντικό το ζήτημα που θα μας απασχολήσει. η πολιτική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζοντας 2020, και το μέλλον βεβαίως της πολιτικής έρευνας να δούμε πού βρισκόμαστε και τι μας περιμένει. Είχε πάρει τεράστια σημασία το πρόγραμμα έρευνας για την Επιτροπή μας διότι είναι η υπεύθυνη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκπόνηση των ε, βασικών της ε, ε, αξώνων και βεβαίως για την παρακολούθηση. Είναι το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για τον ορίζοντα 2020, το επόμενο θα είναι το 9ο είναι δύσκολο να πούμε στρατηγική 2026, δεν θα είναι ίσως τόσο καλή ιδέα να μιλάμε για στρατηγική 2026, διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Προετοιμάζουμε λοιπόν μία έκθεση. Η συγγήτρια είναι η, κυρία Σολεδά Μπεθόν Ρουίθ Ναι, συγγνώμη. Κοίτας αριστερά, ενώ είστε ίσια εδώ στη μέση. Είστε από ό,τι κατάλαβα λοιπόν στο κέντρο, στο επίκεντρο των εργασιών μας. Θα είναι λοιπόν η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενδιάμεση αξιολόγηση του 2020 και βεβαίω θα έχουμε και μια, πρώτο, μια πρώτη εικόνα για το ένατο πρόγραμμα. Η ακρόαση αυτή είναι άλλη μια δραστηριότητα για την προπαρασκευή αυτή τη έκθεση οι ομιλητές στην ακρόαση αυτή έρχονται εδώ, έρχονται εδώ για να μας εμπνεύσουν. Αναμένουμε πολλά από την κοινότητα των, των ερευνητών, αλλά και από τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλοί περιμένουν πολλά από το πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν μιλάμε πια δηλαδή μόνο για τους επιστήμονες, για την ερευνητική κοινότητα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο υλοποίησης. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτές τις προκλήσεις αλλά και τις ελπίδες του 2020. Είναι το μεγαλύτερο ε, πρόγραμμα έρευνα και καινοτομία. μισή ώρε βέβαια δεν αρκούν ε, για να καλύψουμε όλα τα θέματα. Ελπίζω παρόλα αυτά να είναι μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε δύο ενότητες. Θα ήθελα να σας ζητήσω για την πρώτη ενότητα εδώ θα έχουμε τρεις ομιλίες και στη συνέχεια θα γίνει μια συζήτηση. Και στην δεύτερη ενότητα δύο ακόμα ομιλίες και μετά συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συνάδελφο, την κυρία Καμπεθόν Ρουίθ, να κάνει, που θα μας κάνει μια δήλωση. Είστε η συγγήτρια για την Ήτρε σε ό,τι αφορά την έκθεση εφαρμογής, για την εφαρμογή του ορίζοντα 2020, τον να κανείς υπεύθυνος με τέτοια έκθεση, ε, είναι σημαντικό. Θέλουμε να σα δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσετε λοιπόν πρώτοι. Θέλω να στήσω από όλους τους ομιλητές, από και από τους πέντε δηλαδή, μαζί με, και με την εισηγήτρια, να μην ξεπεράσουν τα 12 λεπτά στις παρεμβάσεις τους καλό θα ήταν για να μπορέσει να γίνει και συζήτηση. Λοιπόν, η εισηγήτρια θα αναφερθεί στα κεντρικά ζητήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια βεβαίως θα έχουμε τις ομιλίες και θα έχουμε και κάποιες ερωταπαντήσεις και σχόλια. Παρακαλώ, κυρία θα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι πρόθεσή μου να δώσω κατευθύνσει για την αναθεώρηση του 2020. Μια μικρή εισαγωγή θα κάνω. Το βασικό είναι σήμερα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες, να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί τους. Όπως γνωρίζετε, ε, όσοι συμμετέχουν στην ακρόαση αυτή, Μιλάμε για τη δουλειά που κάνουμε εδώ και κάποιο καιρό. Το, η ακρόαση εγγράφεται δηλαδή στα πλαίσια των εργασιών τη Επιτροπή Ήτρε. Εμεί έχουμε το ρόλο ε, να ασχοληθούμε με την διάμεση αξιολόγηση που θα δώσει κάποιου πολιτικού προσανατολισμού ε, στην ανακοίνωση που θα μα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού 1291 του 2013 του 2020. Η πρόθεσή μα είναι στα πλαίσια τη ακρόαση αυτή. Ε, η ακρόαση εγγράφεται σε μια σειρά από δραστηριότητε, έτσι, έτσι ώστε να συλλέξουν πληροφορίε από όλου τους ε, ενδιαφερομένους φορεί. Θα ήθελα λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω ε, χαιρετώντα σα και λέγοντα σα ε, κάποιοι από του συζητητές είναι εδώ σήμερα ε, και από τι άλλες ομάδες από κοινού γίνεται αυτή η δουλειά. Από το ΕΛΚ είναι η συνάδελφος Μπάρμπαρα Κούμπρικα, από την ECR, η ε, Mambo Suite, από την ALDE, η κυρία Γκέριν και από την Γκουικ Μαρίσα Ματίας η κυρία Μαραγάλο, ο Νταβίτ Μπορέλ, επίσης από την FDD και ο Νικολά Μπέ. Πρόκειται λοιπόν για μια ομαδική προσπάθεια. Θέλουμε λοιπόν να συλλέξουν πληροφορίε από όλου του ενδιαφέροντε φορεί, από την κοινότητα ε, την επιστημονική, τον κλάδο, τον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και ε, τους ίδιους τους θεσμούς για να δούμε πόσο αποτελεσματική και πόσο, ε, πόση συνέπεια διέπει τελικά ε, το πρόγραμμα του 2020 και ποια είναι κυρίως η προσθέμενη αξία αυτού του προγράμματος και ποιος είναι, είναι ο κοινωνικο οικονομικο αντίκτυπος με βάση τους πολιτικούς στόχους που είχαμε θέσει. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε λοιπόν την εφαρμογή και τον αντίκτυπο σημαντικό το θέμα της εφαρμογής, να δούμε πού τα πήγαμε καλά, πού όχι, για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο ένα το πρόγραμμα και ο αντίκτυπος όμως έχει σημασία. Ο αντίκτυπος όχι μόνο οικονομικός αντίκτυπος, διότι γίνεται πολύ λόγος για το οικονομικό αντίκτυπο, το πρόγραμμα Αζόντια 2020 έχει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, πρέπει να εξολογήσουμε όμως και τον αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο συνοχής είναι εξίσου σημαντικό να δούμε δηλαδή πώς βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα αλλά να έχουμε κατά νου ότι ε, η ευημερία των συμπολιτών μας πρέπει να είναι ο βασικός στόχος. Αυτός πρέπει να είναι ο αντίκτυπος. Ανταγωνιστικότητα και συνοχή λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προκλήσεις εγγράφεται όπω ξέρετε στη Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, το ορίζοντα 2020 που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2010. Η καινοτομία και η έρευνα έρχονται στο επίκεντρο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική, όμως η οικονομική κατάσταση, η οικονομική συγκυρία ε, προφανώς ε, ε σημάδεψε τον ορίζοντα 2020. Έχουμε αλλαγέ όμω τώρα, έχουμε εξελίξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτό το μελλοντικό πρόγραμμα το ένα το πρόγραμμα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το όνομά του ακόμα, το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτές είναι οι προκλήσεις. Ε, να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, σε επίπεδο συνοχής και ποιες είναι οι λύσεις, ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες για το επόμενο πρόγραμμα. Ναι. Πλαίσιο. Ευχαριστώ. Μάλιστα να ευχαριστήσω την κυρία Καμπεθανδροήθη για την εισαγωγή της. Πρώτος ο μιλητής ο καθηγητής Αντρέ Μαρτινούτσι από το Ινστιτούτο Διαχείρισης ε, της Βιωσιμότητας και η συγκητής της ε, ε, τη ομάδα εμπειρογνωμόνων αξιολόγηση του 7ου προγράμματος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ασχολείται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με την κοινωνική εταιρική ευθύνη, ε, την έρευνα και την καινοτομία και την αξιολόγησή τους, την υπεύθυνη έρευνα και την καινοτομία. Ε, χρειαζόμαστε και, και αξιολόγηση ex post, αλλά και ex ante και εκ των προτέρων. Ε, για πάνω από 15 χρόνια έχει συντονίσει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο, τα ευρωπαϊκά ταμεία και ε, υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης ε, διαδικτυακό το οποίο έχει θεσπιστεί από τον κύριο Μαρτινούτσι. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία που αναφέρω στο βιογραφικό σας σε συνεργασία με επιχειρηματίες αναλύεται τα ωφέλη αλλά και τις προκλήσεις από την αξιολόγηση αντικτύπου την επιχειρησιακή και τη διαχειρισιακή ε, πώς μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία για την διάχυση της γνώσης Αυτή τη στιγμή συμμετέχετε στην έρευνα για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην, συστήματα συστήματα καινοτομία. Κοινωνία των πολιτών λοιπόν, αλλά και το θέμα της υπεύθυνη καινοτομία έρευνα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία της αποτελεσματική χρήση ε, χρήσης των πόρων στον τομέα της έρευνας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας. Η κυρία Καμπεθάν Ρουίθ εξήγησε την προσέγγισή μας, οπότε ας ξεκινήσει ε, η πρώτη ομιλία. Παρακαλώ κύριε Ματινούτσι. Πρόεδρε Πούζε, κυρία Καμπεσόν Ρουίς, διακεκριμένοι ε, ε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ε, με το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή την ε, κοινωνική πτυχή του προγράμματος Horizon 2000, πώς το μετράμε, αν το μετράμε σωστά και αν μπορούμε να συγκρίνουμε την, ε, τον, το ευρωπαϊκό επίπεδο με τις εθνικές πρακτικές, τι μπορούμε να αποκομίσουμε. Βασίζομαι σε τέσσερις μελέτες που έχουν ήδη γίνει, η εξπόστα αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου υπάρχουν 7 για το οποίο είμαι συγγητής, το ε, σύστημα παρακολούθησης που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια που προσπαθούμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο του 7ου προγράμματος πλαισίου και στι δύο περιπτώσει θα δείτε εκθέσει θα δείτε σύντομα υπομνήματα πολιτική με βάση αυτά τα δύο projects και βασίζομαι και σε άλλε δύο πρόσφατε έρευνε όπου δεν υπάρχουν ακόμα εκθέσει που θα υπάρξουν σε, κάποιε σε λίγες εβδομάδες. Ε, πρόκειται για μια μελέτη για την ανάλυση δικτύου της, ε, των οργανώσεων κοινωνία των πολιτών τα προγράμματα πλαίσια. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος λοιπόν για να αξιολογήσουμε την κοινωνική προσέγγιση. Τότε θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε ολόκληρη τη δομή του Horizon 2000. Γνωρίζετε ότι έχει τρεις πυλώνες το πρόγραμμα. Ε, αυτό μετέτρεψε το FP7 στο Horizon 2020. Ε, μιλάμε για άριστη επιστήμη, βιομηχανική πρωτοπορία και κοινωνικές προκλήσεις. Ε, η λογική του πρώτου που επίσης εντάσσεται στην ε, έρευνα ε, στα πανεπιστήμια που είναι βασικός, ε, η βασική ομάδα στόχος πρόκειται για ανακαλύψεις, για αριστεία και για άτομα όχι, και, όχι ομάδες αλλά άτομα η λογική αυτή του συστήματος είναι η επιστημονική αριστεία που μετράται με δημοσιεύσεις και στα διαδρομίες και επίσης στην διαδικασία που καθοδηγεί ολόκληρο το σύστημα είναι η δημιουργικότητα και η επιλεκτικότητα τα πολύ δημιουργικά μυαλά, υποβάλλουν ευθύ ιδέε, λαμπρέ ιδέε και μετά γίνεται μια διαδικασία επιλογή που βασίζεται σε ε, συμβούλια αξιολόγηση και ε, σε μια ε, προσέγγιση αυτού αυτο, αυτοαξιολόγησης και επιθυμίας. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την εχνηλάτηση των σταδιοδρομιών, υπάρχουν κάποιες παραπλανητικές επιτυχίες, αλλά όταν μιλάμε για κοινωνικό αντίκτυπο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ομάδα των βασικών ερευνητών στην πρωτοπορία συχνά αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο στην κοινωνία ως μια απογοήτευση, γιατί το δικό του στόχο είναι η αριστεία. Φαίνεται να υπάρχει δηλαδή ένα αντιστάθμιο ανάμεσα στην αριστεία από την μια πλευρά και τον αντίκτυπο από την άλλη ειδικά αν δούμε αυτόν τον πυλώνα του Horizon 2020, αν δούμε το δεύτερο πυλώνα, εδώ έχουμε την βιομηχανική ε, πρωτοπορία. Εδώ βλέπουμε ότι ο στόχος είναι οι εταιρείε. Δεν πρόκειται για ανακαλύψεις αλλά για καινοτομία και ο στόχος είναι το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα. Ο οικονομικός αντίκτυπος μετράται με αξιολογήσεις εκ των προτέρων και ε, εκ των υστέρων. Είναι εντυπωσιακό ας πούμε. Η απώλεια θέσεων εργασίας είναι ένας αρνητικός αρνητικός κοινωνικός αντίκτυπος ε, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων συχνά αυτό το σύστημα που βασίζεται στη μεγιστοποίηση του κέρδους δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πάντοτε τις κοινωνικές προκλήσεις. Ένα μικρό παράδειγμα, αντιμετωπίσαμε το θέμα της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικότητας των πόρων. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη ε, δημοσίευσε μια ιεραρχία αποβλήτων. Στόχος είναι να αποφύγουμε τα απόβλητα και όχι να τα μειώσουμε μόνο και αν το εντάξουμε αυτό στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ο, στόχο στόχος δεν, επιτεύ, δεν επιτεύθηκε γιατί μπορεί η βιομηχανία να κερδίσει μέσω της δημιουργίας αποβλήτων και μετά με την πώληση αυτών. Είναι ένας τρόπος να κερδίσουν δηλαδή οι εταιρείε και το να το αποφύγουμε αυτό ε, δεν έχει ε, εμπεδοθεί σε αυτή την περίπτωση, σε, αυτή την, σε αυτό τον τομέα. Τώρα, κοινωνικές ε, προκλήσεις, αν το χρειαζόμαστε, Από αποδομικής άποψης, ναι, επί τη βάση τριών επιχειρημάτων. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει η επιστήμη να έρθει πιο κοντά στον, στον κόσμο. Και αν δεν έχουμε αυτόν τον πυλώνα θα είχαμε την αριστεία Ανακαλύψει, ανακαλύψεις, εφευρέσεις, ε, δηλαδή ερευνητέ και πανεπιστήμια. Μετά θα είχαμε τη βιομηχανική πρωτοπορία που είναι οι εταιρείε. Και εκεί δεν έχουμε καθόλου να κάνουμε με τον κόσμο. Χρειάζεται η προσέγγιση της κοινωνικής πρόκλησης, έτσι ώστε η επιστήμη να έρθει πιο κοντά στον κόσμο και να αντιμετωπίζει θέματα που είναι σημαντικά για αυτόν. Δεύτερο μου επιχείρημα είναι ότι χρειάζεται να δώσουμε λύσεις, να αλλάξουμε πράγματα στον πραγματικό κόσμο και να προωθήσουμε την ευθύνη ως τρίτο στόχο, πέρα από την αριστεία και το κέρδος. Εάν περιορίσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο μόνο στις, ε, στην καινοτομία, στις επιβρέσεις και στο κέρδος ε, και στην αριστεία, δεν έχουμε καθόλου να κάνουμε με τον ε, αντίκτυπο. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε τα καθολικά στοιχεία. Καθολικά στοιχεία γιατί διαφορετικά δεν εντάσσεται πολλοί κόσμο στο πρόγραμμα, ενώ μέσω μιας τέτοιας ε, κοινωνικής πρόκλησης μπορεί αυτό να γίνει με φιλόδοξο και ενδιαφέροντα τρόπο. Τώρα, λειτουργεί αυτό. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση και πώς μετράται η επιτυχία. Με βάση αυτά τα επιχειρήματα, πώς μετράμε την επιτυχία σε σχέση με την προσέγγιση της επιστήμης στον κόσμο και αν λειτουργεί. Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο κόσμος στην επιστήμη. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό επιστημονικά και έχουμε διακρίνει έξι διαφορετικού τρόπου ώστε η επιστήμη να έρθει πιο κοντά στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, ο κόσμο μπορεί να είναι μια ομάδα στόχο για την ενημέρωση και τη διάδοση των πορισμάτων. Οι επιστήμονε κάνουν τη δουλειά του, το ολοκληρώσουν, το δημοσιεύουν και μετά έρχονται σε επαφή με τα μέσα μαζική ενημέρωση και του λένε την ιστορία για το τι ανακάλυψαν. Αυτό πάει καλά στο Horizon 2020. Και όσον αφορά τη διάδοση των ε, επιστημονικών πορισμάτων. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα κίνητρα, αλλά πάντως κατά βάση δουλεύει το σύστημα αυτό. Τώρα, ο κόσμος μπορεί να είναι και μια πηγή στοιχείων. Αυτή είναι η βασική ιδέα των παρατηρητηρίων πολιτών. Δηλαδή δεν συλλέγουν μόνο οι επιστήμονες στοιχεία, αλλά και, ο κόσμος, ε, οι πολίτες. Υπάρχουν κάποια θέματα ιδιωτικού χώρου και όταν μιλάμε για τα μεγάλα δεδομένα big data, εκεί προκύπτει πρόβλημα, πάντως βασικά δουλεύει και αυτό το στοιχείο. Έπειτα, οι πολίτες μπορεί να είναι εταίροι, να έχουμε δηλαδή μια εκπροσώπηση θεσμών, δηλαδή ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να είναι μέρη να εμπλέκονται στα project. Αυτή ήταν μια βασική ιδέα πριν από κάποια χρόνια, να αναμειχθούν δηλαδή οι οργανισμοί τη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Αν δούμε τις μελέτες επί των οποίων έχουμε δουλέψει, το 6% των οργανισμών ήταν των οργανώσεων ήταν ε, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά έλαβαν λιγότερο από 1% της χρηματοδότησης. Ήταν εταίροι αλλά δεν ήταν ε, δικαιούχοι. Είχαμε 80% εγκατάλειψη ε, των προγραμμάτων από το πρόγραμμα πλαίσιο 6 μέχρι το πρόγραμμα πλαίσιο 7, στη μετάβαση δηλαδή. Ε, δηλαδή οι οργανώσει της κοινωνίας των πολιτών εγκατέλειψαν τα προγράμματα, είναι στην περιφέρεια των δικτύων, ενώ οι μικρομεσαίε επίση σταμάτησαν να ασχολούνται κατά 70%. Η συμμετοχή λοιπόν τη Κοινωνία των πολιτών ω εταίρου δεν λειτουργεί γιατί έχουν διαφορετική λογική, του ενδιαφέρει περισσότερο αντίκτυπο παρά τα απορίσματα τα ερευνητικά και θέλουν περισσότερο, ενδιαφέρονται περισσότερο για τι πολιτιστικέ διαφορέ. τρία ακόμα στοιχεία που δεν εφαρμόζονται μέσω του προγράμματος του πλαισίου. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τα συμβούλια ηθικής σε επίπεδο project και προγράμματος, οι, οι, οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών, οι οργανώσεις, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φύλακες, ως οργανώσεις ελέγχου και να κάνουν δηλαδή έρευνες και προτάσεις ε, που αυτή τη στιγμή γίνονται από τους ίδιους τους ερευνητές ε, και οι ε, αξιολογήσεις αντικτύπου επίσης από τους ερευνητές. Θα ήταν εύκολο να συμμετέχουν εκεί οι οργανώσεις των πολιτών, τουλάχιστον για το ε, πτυχή του αντικτύπου και έπειτα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για την θέσπιση της, των, της θεματολογίας ε, που είναι μια διαφανής διαδικασία μέχρι στιγμής και υπάρχει πολλή γνώση, ε, θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα που θα ονομάζεται οράματα και θεματολόγια, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Αυτά λοιπόν για το κατά πόσο η επιστήμη πάει πιο κοντά στον κόσμο. Τώρα, παροχή λύσεων. Αν και δεν είναι γραμμικό το μοντέλο, ε, περνάει καιρό από την εφεύρεση στην καινοτομία, γιατί πρέπει να πάει ε, περάσει διάφορες φάσεις. Ανακαλύψει ένα φαινόμενο, θεωρία ε, και μετά αυτές οι θεωρίες οδηγούν σε τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγικές. Εκεί εντάσσεται ο επιχειρηματικός τομέας και μετά εξαρτάται από τους αγορές και από τους εάν θα προτιμήσουν αυτό το νέα προϊόντα ή τις νέες υπηρεσίες και στο τέλος πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο. Στο τέλος λοιπόν έχουν περάσει 5 με 20 χρόνια. Αν θέλεις λοιπόν να δεις αν η λειτουργία της, κοινων... της... της προσέγγισης ε, προκλήσεις κοινωνικές ε, λειτουργήσε, παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δεν περιμένουμε λοιπόν τεράστια συμβολή εξ αλλά μπορούμε να τα κρίνουμε εξάντε και αυτό κάναμε με αυτό το σύστημα παρακολούθησης. Έχουμε εκ των προτέρων εκτιμήσει τη δυνητική συμβολή που μπορεί να έχει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους αυτή που έχουν θεσπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο πριν από λίγους μήνες, όπου σχεδόν 200 χώρες υιοθέτησαν αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τώρα είναι και η και η ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2030. Ε, άρα λοιπόν δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχεία με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά με τα θέματα αυτής, ας πούμε, για την υγιή ζωή, ε, για την ενέργεια και για την βιώσιμη κατανάλωση έχει υπάρξει αντίκτυπος 60% των project και περίπου τα 3 τέταρτα της Ευρωπαϊκής Συμβολής ε, πήγε σε προγράμματα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο για την επίτευξη των στόχων ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν είναι εξπόστη γιατί είναι πολύ νωρίς, αλλά ε, τα πορίσματα είναι πολύ αισιόδοξα σε σχέση με τον πιθανό αντίκτυπο. Τώρα, πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα, τα στοιχεία καθολικότητας στο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα οι τρεις πυλώνες είναι χωριστοί. Αν θέλουμε να είναι πιο καθολικοί, θα πρέπει να σχεδιάσουμε συγκεκριμένους χώρους για την ε, συμπαραγωγή γνώσης και καινοτομίας, καθώς και να να μίξουμε, να εμπλέξουμε πολλούς και διάφορους ε, φορείς, καθώς και να μιλήσουμε για τοπία και όχι για projects. ώστε να αναπτύξουμε λογικές παρέμβασεις. Τελευταία ερώτηση αφορούσε εθνικά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά εθνικά παραδείγματα. Θα χρειαζόμουν δυόμιση ώρες, τρεις ώρες για να σας δώσω παραδείγματα. Αν υπάρχει προστιθέμενη αξία, πιστεύω είναι πιο σημαντική ερώτηση. Προστιθέμενη αξία για το ότι η Ευρώπη ασχολείται με αυτά τα θέματα ή μήπως θα έπρεπε να τα αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Εγώ θα έλεγα ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εξαρτάται από τον τομέα και καινοτομίας για τον οποίο συζητάμε. Αναλόγω με την τεχνολογία, τον τομέα, την πρακτική, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Υπάρχουν ερευνητικοί τομεί με μεγάλε επενδύσει, στι υποδομέ, αλλά και ερευνητικέ ε, ε, δραστηριότητε που είναι πιο οριζόντιε. Η πιο σημαντική προστιθέμενη αξία είναι η απλοποίηση, η πρόσβαση στα στοιχεία και η δημιουργία θεματολογίου. Είναι σωστό, ναι. Να διατηρήσουμε τους τρεις πυλώνες χωριστά, θα πρότεινα να μην συγχωνευτεί η έρευνα με στόχο την ε, έρευνα, ε, με να έρθει η επιστήμη πιο κοντά στον κόσμο, να συνδεθούν ε, το πρόγραμμα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να αναπτύξουμε τομείς και όχι να συνεχίσουμε με τη μικροδιαχείριση μικρών projects. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, προσέγγιση κοινωνική πρόκληση υπό το ορίζον 2000. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. βεβαίω ε, όλα τα ε, ερωτήματα και τις παρατηρήσεις σας για το πώς μετράμε τον αντίκτυπο ή τις εθνικές καλές πρακτικές, τα παραδείγματα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας και σας ευχαριστώ για την εισηγησή σα και τώρα περνάμε στην στο επόμενο, θέμα, στην Εν γέννη πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Πολιτική καινοτομία και όχι μόνο για την έρευνα και με μονομένους δικαιούχους έναντι προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ πολλών δικαιούχων. Ίσως και αυτή η ιδέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καινοτομία είναι καλή. είναι ενδιαφέρον να δούμε κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Και τώρα η κυρία Ζόνενφέλντ. Από το Ευρωπαϊκό Σωτό της, ε, του Πανεπιστημίου της Γάνδης. Όχι. Ε, από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ Λογοτεχνία και Γλώσσες, ε, σύμβουλος πολιτικής ε, για την έρευνα στη Γάνδη και εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. και στο, στα ευρωπαϊκά όργανα. και σχέσεις στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας με τους εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα θεσμικά όργανα ώστε να έχουν μια αποτελεσματική συνεργασία. Υποστηρίζετε το ΕΡΑ και έχετε επίσης την ευθύνη της διάσκεψης των Britannian Flamdems και της ανανέωσης της έρευνας. Είστε πρόεδρος του κοινού προγράμματος έρευνας του Διαπανεπιστημιακού Ερευνητικού Συμβουλίου με ιδιαίτερη έμφαση πρόσφατα στις κοινωνικές επιστήμες και τον ορίζοντα 2020. Όλα αυτά πολύ ωραία, απλώς για μας η πιο σημαντική ε, συμβολή θα ήταν η ε, ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καινοτομία που έχουμε στο εγγύς Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την παρουσίαση και ευχαριστώ την κυρία Καμπεσόν Ρουίς για την παρουσίαση. Πρώτα θα ήθελα να εξηγήσω το δικό μου πανεπιστήμιο τι κάνει πριν περάσω στο ΕΑΣΥ είναι στην παρακολούθηση της υλοποίησης του 2020 με το έγκλο. Είμαστε μέλος της EUA και της ΕΖΑΡ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει πρώτο καθεδρία στην έρευνα SSH. Ας δούμε όμως τι είναι το EIC. Όταν αρχίσαμε να προετοιμάζουμε αυτήν την ε, συνεδρίαση πληροφορίες πολλές από το EIC δεν υπήρχαν. Αλλά νομίζω ότι τώρα μπορούμε να το περιγράψουμε ως έρευνα στηριζόμενη στις ανάγκες της αγοράς. Με βάση τη ζήτηση δηλαδή. Έχουμε ένα είδος υπηρεσίας μεταφοράς τεχνολογίας και αυτό εξυπηρετεί και τους φοιτητές μας συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το EIC ε και μας ενδιαφέρει η διασύνδεση μεταξύ του EIC ε και των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Προϋπολογισμός. Ο κύριος Γιουνκέρ στην ομιλία για την κατάσταση Ένωση το Σεπτέμβριο μας είπε ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο προϋπολογισμός της έρευνας προς όφελος του EIC. Αν με συγχωρείτε γιατί ξεχνάω και τις διαφάνειες. Ο προπολογισμό ήδη έχει ξεφύγει από το ορίζον και έχει περάσει στο έτσε. Το έτσε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για μας ιδιαίτερα στηρίζεται στην καινοτομία. Άρα πρόκειται για ένα είδος δανεισμού από την έρευνα στην ε, πανεπιστημιακή κοινότητα. Εμείς θα θέλαμε να επανέλθουν τα κονδύλια που έχουν περικοπτεί από το ορίζον ε, προς χάρη του έτσε. Μας έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα αυτές οι περικοπές. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας προσφέρει στις αιτήσεις διαδικασίε για τον προπολογισμό εναντί των περικοπών. Σας ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε να συνεχίσετε και να αποτρέψετε άλλες περικοπές στον προπολογισμό της έρευνας. Επίσης θα θέλαμε, απευθυνόμενοι στους υπουργούς των οικονομικών σας, της χώρας σας, να επιδιώξετε μία λύση προς την κατεύθυνση των επενδύσεων και όχι τόσο στην περικοπή του κόστους. Κάτι ακόμη. Τα πανεπιστήμια στηρίζονται σε χορηγίες. Δεν παράγουμε, δεν πουλάμε τίποτα. Δεν παράγουμε έσοδα, δεν έχουμε κέρδος. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να επιστρέψουμε δάνειο. Το έτσι λοιπόν έχει πάρει χρήματα της καινοτομίας. Αν δείτε όμως τα προγράμματα πλαίσιο, και θα το πω πολύ απλά, τα προγράμματα πλαίσιο 6 και 7 μιλούσαν ιδιαίτερα για την έρευνα, το Horizon για την καινοτομία. Έχει έρθει η ώρα τώρα νομίζω να εξισορροπηθούν οι δύο αυτές προσεγγίσεις και ελπίζω να μας βοηθήσει αυτό το Κοινοβούλιο. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στην έρευνα και καλύτερα να εξορροπηθεί η θέση της στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα ιδιαίτερος. Μια σύσταση θα θέλαμε να απευθύνουμε κατά τρόπο ξεκάθαρο και πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο για σας να υποστηρίξετε τις ερευνητικές δραστηριότητες έχουμε τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας και στο δεύτερο πυλώνα και στο τρίτο. Αλλά ε, έρευνα μόνο δεν υπάρχει πουθενά. Καινοτομία μόνο υπάρχει, αλλά όχι έρευνα. Για να υπάρχει λοιπόν μέσα στο ορίζοντα, στο 2020 ιδιαίτερα η μνήμα στην έρευνα, πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για ερευνητικά μόνο προγράμματα. Γιατί και για καλύτερη εξισορρόπηση των δύο στοιχείων, των δύο σκελών, έρευνας και ε, αλλά και, και γιατί η εισαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ενοποίηση SSH, η οποία σχετίζεται ιδιαίτερως με τους προσανατολισμούς που θα δώσουν οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα. Η πολυτομεακή προσέγγιση του ορίζων ήταν καλή, αλλά μέχρι ενός βαθμού. Επίσης, συστάσεις της DGRTD, Network Analysis, καταγράφουν ότι η υπερβολική προσέγγιση διατομεακή μπορεί να έχει αντίξωη συνέπεια στην καινοτομία. Και επίσης η αναγκαιότητα από ό,τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το FED Open να μετακινηθεί στο EIC. Πράγμα το οποίο για μας μπορεί να δημιουργήσει ε, προβλήματα γιατί μέχρι τώρα αυτό προσέφερε δυνατότητες για έρευνα ανακαλύψεων ή εφευρές ανακαλύψεων. Ε, αν όμως μετακινηθεί δεν θα μπορέσει να αφήσει περιθώριο για δραστηριότητα ανακαλύψεων. Συζητήσεις έχουν γίνει εδώ στις Βρυξέλλες για την ε, χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων είτε προς ένα μόνο φορέα είτε συνεργατικών. Εμείς θέλουμε και τα δύο να υποστηριχθούν. Ε, τα πρώτα επιτρέπουν την ευρωπαϊκή υπεροχή, την ευρωπαϊκή προστομένη αξία, ενώ η συνεργατική δράση είναι απαραίτητη όταν άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη αυτό και ίσως θα ήταν σκόπιμο να εξετάσετε δυνατότητες για πιο στενή συνεργασία σε εθνικό και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά με ιδιαίτερο μέλημα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, ώστε να υπάρχουν κανόνες NEA, ε, οι κανόνες του ορίζον, και να μην δημιουργηθούν και άλλα προγράμματα γύρω από αυτό που δεν θα συνιστούσαν βέβαια απλοποίηση. Περισσότερη ενοποίηση λοιπόν στον ερευνητικό κλάδο στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει και ένα χάσμα έρευνας και καινοτομίας. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει στην ε, Γάνδη και σημειώνουμε όταν η Επιτροπή λέει ότι δεν είναι ταμείο συνοχή στο ορίζον, ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το κενό αυτό μεταξύ έρευνα και τεχνολογίας. Το ορίζον είναι μια πολιτική που συνοδεύει την έρευνα και η καινοτομία, όπως λέει η Επιτροπή, και σε αυτό την υποστηρίζουμε. Πρέπει όμως και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως κάνουμε και εμείς στη Γάνδη με το SIP, με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Ας παραμένει λοιπόν αυτή η δυνατότητα για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση. Μπορεί να βελτιωθεί το Sea of Excellence Scheme. Πρόσφατα μάλιστα Αναφέρθηκε από την Επιτροπή ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερω. Συνεργατικέ σχέσεις επίσης, αρθρωτικά ταμεία και ορίζον δηλαδή, όπου όμως κρίσιμη σημασία θα έχει αυτές οι συνεργατικέ σχέσεις να αναπτυχθούν σε επίπεδο προγραμματικό, στρατηγικό. Γιατί βλέπουμε από την εμπειρία μα και από την έρευνά μα στο Πανεπιστήμιο τη Γκάνδη ότι είναι πολλές οι διαφορές στην ορολογία μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Πολλά είναι τα στοιχεία που δεν είναι ευθυγραμμισμένα όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, Φερρυπίν. Τα λογιστικά συστήματα, τα συστήματα λογοδοσίας. Δεν είναι λοιπόν εύκολη υπόθεση αυτή η ανάπτυξη συνεργασιών. Μπορούν να απλουστευτούν περισσότερο. Για μας καλή ιδέα δεν συνιστά το να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός για την δικτύωση και τα ταξίδια του ορίζουν για να κλείσει όπως λέγεται το κενό έρευνας και καινοτομίες υπάρχουν ούτως ή άλλως το έρανε, το CSA και άλλα μέσα αλλά πρέπει αυτοί οι προϋπολογισμοί να αξιοποιηθούν για, το, για την κάλυψη του κενού έρευνας και κοινολογίας όπως Άλλωστε είναι και ο στόχος του ορίζον. Όπως είπα και νωρίτερα, το Πανεπιστήμιο της Γάνδη έχει την πρωτοπορία στην συνεργατική έρευνα SSH. Αναζητά έρευνες από όλη την Ευρώπη, διαδικασίες συνοδείας με παρουσία ε, συνεργατών SSH που όμως δεν μπορεί να μετατραπεί πάντοτε σε πολυτομεακή συνεργασία. Η Επιτροπή μας λέει ότι είναι μια πολύ μακρά διαδικασία αυτή του SSH. Εφόσον θεωρούμε θα πρώτα πόρη μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Όσον αφορά τις συστάσεις από πλευράς μας, ιδιαίτερη σημασία έχει η ποιότητα Δεν θυμάμαι κανέναν επιστήμονα να μου λέει ότι από πω κατάφερα κάτι συγκεκριμένο από τη μια μέρα στην άλλη χάρη σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρόκειται για συνεργασίες και σε αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στον ορίζοντα. Ίσως ένας προπολογισμό συγκεκριμένο θα μπορούσε να προβλεφθεί για τα υφιστάμενα KPI και την έκθεση παρακολούθησης του SSH KPI γιατί λοιπόν, εάν θέλουμε πράγματι να κοιτάξουμε αυτό το θέμα, ίσως θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ένα συγκεκριμένο προπολογισμό. Επίσης, ε, το συνεργατικό έργο για τις καινοτόμες μικρομεσαίες θα μπορούσε να ανοίξει και σε, μικρο... και σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, γιατί τίνει να είναι κλειστό σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να αφορά μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν γίνει αυτό θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την κοινωνική καινοτομία. Και επίσης, οι ερευνητικές δράσεις έχουν βελτιώσει την ποιότητα του ΙΣΙΑ. Αναφέρθηκε ήδη. Εμείς υποστηρίζουμε το έγκλο της συστάσεις και χωρίς να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, το SSH ως ιδιαίτερη αξία και νομίζω ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει να ενσωματώσει την ε, έρευνα του SSH στην, ε, στις εκθέσεις της. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουμε ότι προσδιορίζει καλύτερα τις, ε, την αξιολόγηση συνεπειών. Ιδιαίτερα για τους ερευνητές SSH που δεν είναι τεχνικοί ερευνητές, ερευνητές τεχνολογίες. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αέρα και τον δημοσιονομικό κανονισμό και την απλοποίηση. Οι προτάσεις και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του ορίζων έχουν όλο και περισσότερα τετραγωνίδια που καλείται να ε, συμπληρώσει προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη για το αέρα. Βεβαίως δεν είναι κακό το αέρα αλλά τα τετραγωνίδια θα μπορούσαν να καλύπτονται σε θεσμικό επίπεδο. Η πολιτική ολοκληρωμένη έρευνα, σε παραδείγματι, η, το, η σήμανση υπεροχής HR είναι κάτι που μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει μαζί με τα layers σε θεσμικό επίπεδο μπορεί τα τετραγωνίδια δηλαδή να τα συμπληρώνει, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τον ερευνητή και την ε, μονάδα υποστήριξη έρευνα. Και μια τελευταία παρατήρηση εδώ για το δημοσιονομικό κανονισμό. Η Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού αυτή τη στιγμή και όχι έρευνα προτείνει Ε, χρηματοδότηση στηριζόμενη σε αποτελέσματα. Εμεί όμω ω ερευνητικό, ω πανεπιστήμιο, δεν, δεν, δεν μπορούμε να δεχθούμε χρηματοδότηση με βάση αποζημίωση στηριζόμενη σε αποτελέσματα. Θα προτείναμε λοιπόν άλλο σύστημα, πιο απλό, αποζημίωση δαπανών, επί παραδείγματι. Για μας. Που δεν γνωρίζουμε ε, ποιος εφήβρε τον όρο απλουστευμένα πρότυπα κόστους, γιατί αντιθέτως από απλούστευση μάλλον περιπλέκουν την κατάσταση, πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα απλουστευμένα πρότυπα κόστους και άλλοι τύποι αξιολόγησης όπως ε, βραβεία, κόστος αναμονάδα, κλινικές δοκιμές. Ίσως μπορούν να προσφέρονται για ενοποιημένα προστευμένα συστήματα απολογισμού κόστους αλλά όχι για κάθε τύπο έρευνας. Γι' αυτό παρακαλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη που προβλέπει η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών. Ευχαριστώ πολύ τώρα η κυρία Καμπεθόν Ρουίς έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον πρώτο ομιλητή κυρίως. Έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα, το είπα και εγώ στην εισαγωγή μου γενικότερα, την αναγκαιότητα λοιπόν η επιστήμη να βάλει τον πολίτη στο κέντρο της του όλου εγχειρήματο να απευθύνεται στον πολίτη. Νομίζω ότι οι κοινωνικές επιστήμες και ο κοινωνικός αντίκτυπος ε, της έρευνας είναι κρίσιμος. Έγινε αναφορά στην αξιολόγηση βέβαια, το πώς μετράμε αυτόν τον αντίκτυπο. Το ερώτημά μου είναι πώς, ε, ποιο είναι το κριτήριο όταν γίνεται μια αξιολόγηση των διαφορών προγραμμάτων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση την κοινωνική. Να το εξηγήσω κάπως. Δώσατε το παράδειγμα ε, της απώλειας ε, της θέσης εργασίας ε, λόγω της τεχνολογικής προόδου ως δηλαδή αποτέλεσμα της έρευνας ουσιαστικά και της επιστημονικής πρόοδου. Θα ήταν καλό να υπάρχει ένας τρόπος να το μετρήσουμε αυτό οριζόντια εκ των προτέρων έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι προκλήσεις που εμφανίζονται από την ίδια την καινοτομία και την έρευνα. Και για την εκπρόσωπο της, ε, την καθηγήτρια μάλλον του Πανεπιστημίου της Γάνδης, ε, αναφέρθηκαν πολλά ζητήματα, πολλές προκλήσεις που πρέπει να δεχθούν υπόψη στην καρδιά και της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ η ομιλήτρια. Είναι δύσκολο να συμμετάσχουν κάποιοι, κάποιοι οργανισμοί. Ε, αυξάνονται τα δάνεια, μειώνονται οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Δεν θέλαμε λοιπόν περισσότερες εξηγήσει από αυτού. Ε, τι πιστεύετε εσείς, σε περιπτώσει, πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τον ένα τον άλλο τομέα το να περάσουμε από τις ε, ε, ενισχύσεις στα δάνεια στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Και βεβαίως το θέμα της αξιολόγησης ε, των, με βάση τα αποτελέσματα. Εάν χρηματοδοτήσουμε με βάση τα αποτελέσματα, πώς θα το μετρήσουμε μετά. Αυτό πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση εξάντε. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Ε, Ευχαριστώ. Να ακούσουμε ακόμα μερικά ερωτήματα όμως. Η κυρία Κουντρίσκα από το ΕΛΚ σκιώδης εισηγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τις παρουσιάσεις, επίσης αυτές τις ομιλίες. Ε, ε, πραγματικά μαθαίνουμε πολλά με τέτοιου είδους ε, παρουσιάσει να ευχαριστήσω την κυρία Καμπεθόν Ρουίθ για την, πολύ ενδιαφέρουσα προποστολή ε, την επίσκεψή μας στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, όπου είδαμε προσώπους ε, της επιστημονικής κοινότητας, ε, καθώς και Πριτάνης από την Ισπανία, την Πορτογαλία. Είχαμε έτσι την αξιολόγηση τη δική τους του ορίζοντα 2020. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γιατί, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του προγράμματος πλαισίου, ποιος είναι ο υποτιθέμενος σκοπός. Εάν επικεντρωθούμε μόνο στις προτάσεις που ακούσαμε από την ε, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γάντης, ναι εντάξει αυτό το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, εάν θέλουμε όμως να αναπτύξουμε ένα νέο πρόγραμμα πλαίσιο, και αν θέλουμε να γίνει μια καλή αναφορά ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια καλή έκθεση με βάση την εμπειρία του ορίζοντα 2020, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποια θα είναι η βάση του νέου προγράμματος και κατά πόσο ο σκοπός είναι όντως ε, να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες για όλους και να συμπεριληφθούν τελικά και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Εμένα μου αρέσει ο τρόπο που χρηματοδοτούνται αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα ταμεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό, όπως το Ταμείο Συνοχής. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αυξάνει το ΑΕΠ της, αλλά, που θα, αλλά να μπορεί να είναι και ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες ε, οικονομίες αναπτυσσόμενες, όχι μόνο ε, τις ΗΠΑ αλλά και την ε, Κίνα, την Ινδία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όταν διθέτουμε χρήματα στην έρευνα τι πρέπει να αφιερωθεί στην βασική έρευνα, τι πρέπει να αφιερωθεί στις ανθρώπινες επιστήμες. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου η αριστεία ε, και η ποιότητα της έρευνας ε, θα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο είναι πολλοί ερευνητές ε, οι οποίοι ως τώρα δεν έχουν πρόσβαση στις υποτροφίες, ε, να φροντίσουμε να έχουν αυτή την πρόσβαση, να μειώσουμε τις τοπικές, τις περιφερειακές ανισότητες και η, αυξημένη ποιότητα της έρευνας να είναι παρούσα σε ολόκληρη την Ένωση και όχι μόνο σε μέρος της Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό, διότι εκεί βασίζεται η όλη φιλοσοφία του επόμενο πρόγραμμα του πλαισίου. Εάν δούμε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την κοινοτομία, το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα των ε, ταμείων συνοχής, ε, εκεί θα δούμε ότι απομακρυνόμαστε τελικά από το στόχο μας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και τώρα η κυρία Λιμπάτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι ανησυχίες που εμφανίζονται στο το 2020 πριν πάμε προς ένα νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις σας και οι δύο σας αναφερθήκατε σε κάποια project τα οποία εφαρμόζονται σε αυτά τα προγράμματα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω γιατί σε κάποιους τομείς είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά επιτυχίας. Δεν μπορώ να βρω μια απάντηση και στο εξής ερώτημα. Γιατί υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη ε, και την αποτελεσματικότητα κατά την υλοποίηση ε, ή κατά, την, ε, κατά τα κατά την υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες. Αυτά είναι εμπόδια που δεν έχουν να κάνουν με την έλλειψη ανθρώπινων πόρων έχουν να κάνουν ενδεχομένω με το γεγονό ότι το κεφάλαιο είναι πολύ κατακαιρματισμένο ή μπορεί να μην υπάρχει επαρκή παράδοση συνεργασία μεταξύ τη επιστημονική κοινότητα και των επιχειρήσεων. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα εμπόδια και πρέπει να τα εντοπίσουμε για να καταλάβουμε γιατί τελικά κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση. Κάτι άλλο που έχει σημασία σε αυτό που είπατε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια τυπικά εμπόδια που δεν μας επιτρέπουν να υπάρχει πλήρη συνέργεια μεταξύ των διαθροντικών ταμείων και του ορίζοντα 2020. Όμως η έλλειψη συνέργειας σημαίνει ότι τελικά πετάμε λεπτά, λεφτά από το παράθυρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα κέντρο έρευνας ε, για συγκεκριμένες θεραπείες. Ε, είναι ένα κέντρο έρευνας αφενός, αλλά από την άλλη ε, εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Ε, θα πρέπει να χρηματοδοτείται και από τα δύο ταμεία λοιπόν. Όταν θα κάνουμε λοιπόν την αναθεώρηση, θα κάνουμε πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να διευκολύνουμε τι συνέργειε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Για του πράσινου τώρα ο κ. Μαραγκάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ακούστε, Νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά το ρόλο και την πολιτική της Ένωσης ξεκινώντας από αυτό που ουσιαστικά είναι και το συμπέρασμα εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα εξαιρετικά ισχυρό, έτσι, εξαιρετικά μεγάλο. Προέρχεται από τα προηγούμενα προγράμματα, το 7 πρόγραμμα πλαίσιο κτλ. Αλλά εδώ φαίνεται και ανεπάρκεια σε περιεχόμενο ε, πολιτικής. Αυτό νομίζω πως είναι στο επίκεντρο ε, της προσπάθειας ε, εξέβρεσης ισορροπιών. Και σήμερα το, το βλέπουμε και στις αποστολές που πάμε ε, αριστεία, ανταγωνιστικότητα, συνοχή, χρειάζεται ισορροπία και δεν έχουν φτάσει στην ισορροπία αυτή. Αφενός τα αποτελέσματα πρέπει να τροφοδοτήσουν την ε, σύγκληση μεταξύ των διαφόρων χωρών ε, αφετέρου όμως τελικά εφόσον δίνουμε έμφαση στην αριστεία και στην ανταγωνιστικότητα τελικά μεγαλώνει το χάσμα καταλήγουμε να βοηθάμε αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν πλεονέκτημα οι οποίοι ήδη έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες αριστείας η ισορροπία μεταξύ των πόρων που διατίθενται και το ποσοστό επιτυχίας. Δηλαδή η επιτυχία των διαγωνισμών είναι η αποτυχία του προγράμματος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες του προγράμματος. Η, η, ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και έρευνας. Εντάξει υπάρχει ένα τεχνολογικό κενό. Αλλά στην αρχή του 2020 όταν τελείωσε η προηγούμενη περίοδος είχαμε πει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τεχνολογικό κενό, το τεχνολογικό χάσμα. Όμως ε, τελικά η βασική έρευνα ε, ουσιαστικά αφέθηκε και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε από ότι στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αφέθηκε στη μοίρα τη. Δίνεται έρευνα στην ανταγωνιστικότητα και στην αριστεία, αλλά αυτό έχει επιπτώσεις και στους το πώς οι πόροι διατίθεται στον ένα ή τον άλλο κλάδο. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα επίλυση στον τομέα της υγείας. Ε, εκεί χρειάζεται έρευνα, βασική έρευνα, έρευνα με κοινωνικούς ε, ε, σκοπούς, όχι με σκοπούς άμεσης οικονομικής απόδοσης. Βεβαίως υπάρχουν κάποια σημαντικά project στον τομέα της υγείας, αλλά η καταπολέμηση των ε, ασθενειών, ε, της άνοιας, ε, του διαβήτη, ε, μια σειρά ασθενειών όπως το AIDS, αυτή είναι κάπως είναι χαμένη κατά κάποιο τρόπο του νέου προγράμματος. Και κάτι ακόμα, Πρόεδρε, και τελειώνω. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι εξαιρετικά ισχυρό, αλλά αντί να συμπληρώνει ε, τα εθνικά προγράμματα, τα υποκαθιστά, ειδικά σε εποχή κρίσης. Και κάποιες χώρες ε, βολεύονται με αυτό. Κάνουν περικοπές στα δικό τους προγράμματα, γιατί ξέρουν, θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα επιλύσει το πρόβλημά τους. Πρέπει να καθορίσουμε προτεραιότητες ε, και πρέπει να πάρουμε και ρίσκα για να κάνουμε πραγματική πολιτική. Ε, κοινωνική προτεραιότητα και να βρούμε τις κατάλληλες ισορροπίε λαμβάνοντα υπόψη την βασική έρευνα. Μάλιστα, ε, πολύ ενδιαφέροντα, όλα αυτά, αλλά υπάρχει ένα όριο. Η κυρία Βιέρνικ, η σκιώδη εισηγήτρια από την Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τους ε, δύο μελετές που μας έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Από τη πλευρά του ΑΛΤΕ, εμείς ξεκινάμε από την ε, αρχή ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα πρέπει να διατηρήσει τις βασικές αρχές του που είναι πολύ σημαντικές ε, για την έρευνα και για την Ευρώπη. Πρέπει να τονίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, σε σχέση με τις μεγάλες βιομηχανικές ε, ε, δυνάμεις και το δίκτυο 2020 παίζει, σημαντικ... παίζει θεμελιώδη ρόλο. Η προηγούμενη έκθεση ανέφερε διάφορα κρατημέλη που τίνουν να αντικαθιστούν την έρευνά τους από το πρόγραμμα ε, ορίζουν 2020. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη στήριξη την, ε, της έρευνας μέσω κονδυλίων ή άλλων μέσων που ε, δεν θα απορρέουν αυτόματα από το πρόγραμμα 2020, αλλά από το κάθε κράτος μέλος, για να τονίσουμε το ενδιαφέρον της έρευνας. Και να θέσω και μια ερώτηση στον τελευταίο μιλητή, τελευταία μιλήτρια. Μιλήσατε για τη χρηματοδότηση διαφόρων τομέων ή και ε, τοπίων σε σχέση με άλλα προγράμματα. Τι, τι εννοείτε, μιλάτε για ευρύτερε πρωτοβουλίε ή αντίθετα για πιο μικρές πρωτοβουλίες. Δεν κατάλαβα, ομολογώ, τον όρο που χρησιμοποιήσατε landscape τοπία. Ευχαριστώ και θυμίζω ότι για τις συνεργασίες θα έχουμε το επόμενο θέμα. Νέες προκλήσεις όπως μετανα... και η τέταρτη ενότητα αφορά το, τις νέες προκλήσεις όπως τη μετανάστευση και άλλα στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 9. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Σε παρακαλώ τώρα να μας δώσετε, αν μπορείτε, απαντήσεις. Μάλιστα. Ε, να πω πρώτα γενικά, αν το πρόγραμμα πλαίσιο αντιμετωπίζει τα όσα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πρώτη ερώτηση και ενδιαφέρεται μόνο για την ανταγωνιστικότητα ή μόνο ή και για θέματα πολιτικής. Και ποια θέματα πολιτικής αντιμετωπίζει το ορίζον 2020. Αν δούμε πιο στενά τον πυλώνα των κοινωνικών προκλήσεων, ε, να δούμε αν αντιμετωπίζει τα ε, ε, προβλήματα. Ποιο θέμα είδε τη μεγαλύτερη αύξηση. Υγεία, όχι. Οι κλιματικές αλλαγές, όχι. Κινητικότητα, Ναι. Οι Ευρωπαίοι για αυτό το θέμα ενδιαφέρονται, την κινητικότητα. Αυτή είναι η πρόκληση που θέλει να αντιμετωπίσει, θέλουν να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή πολιτική. Το πρόβλημα του το μεγαλύτερο είναι η συμφόρηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προβληματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, η κοινωνία των πολιτών είναι, ενσωμα... είναι ε, ενσωματωμένη και δεν πρόκειται για τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Όχι. Το θέμα είναι πώς έχουν να σωματωθεί, ε, ε ομάδε στόχο ή παίζουν και κάποιο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Για την ώρα όχι, δεν έχουν τέτοιο ρόλο. Αν θέλετε λοιπόν να είναι πιο κοντά στον κόσμο θα πρέπει να του αναθέσουμε συγκεκριμένο ρόλο. Άμα θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο Επίτροπος Μοέδας, θα πρέπει να το ανοίξουμε στον κόσμο. Και όταν μιλάμε για προγράμματα χρηματοδότησης, να δούμε ε, πώς λειτουργεί το Horizon 2020 σε σχέση με τις κρατικές, τα κρατικά έργα, όπως ας πούμε κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου. Ας πούμε, από τη Βιέννη στην Πράγα δεν υπάρχει αυτοκινητόδρομος. Ξέρεις που πρέπει να ξεκινήσεις, που πρέπει να πας, ξέρεις ποια είναι τα τοπογραφικά στοιχεία και μετά συνδυάζει διάφορα χωράφια και χτίζεις τον αυτοκινητόδρομο. Και ακριβώς έτσι λειτουργεί αυτό το θέμα των κοινωνικών προκλήσεων. Όμως η ισοκοινωνία έχει μια σταθερή τοπογραφία ή αλλάζουν οι στόχοι. Μήπως είναι κάτι πιο δυναμικό. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Τα μικρότερα ζητήματα είναι ποια είναι η λογική. Αν δηλαδή εμεί απλά δίνουμε αποτελέσματα, και αυτό είναι ο ρόλο τη κοινωνία, να έχουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο που δίνει αποτελέσματα και αν δίνει αποτελέσματα αποκλείουμε τον κόσμο. Εντάξει, άμα αποδίδουμε δηλαδή, φτιάχνουμε θέσει απασχόληση, θέλουμε να έχουμε τεχνολογίε, α πούμε θεραπεύουμε τον καρκίνο, δεν χρειάζεται να εντάξουμε τον κόσμο γιατί έχουμε απόδοση. Αυτό μπορεί να είναι μία άποψη. Τελικά όμως ο κόσμος μπορεί να μην ενδιαφέρεται. Θέλουμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες, γι' αυτό μίλησα για ε, τεχνολογικά τοπία. Ε, τοπία τεχνολογικά, όχι ε, φυσικά. Τώρα, για τις επιτυχίες υπάρχει και τους παράγοντες επιτυχίες, κρατούν κάποιοι μύθοι, θα πρέπει να δούμε τους τομείς όπου οι προτάσεις ξεπερνούν τα κατόφλια. Αν έχουμε ένα ελάχιστο κατόφλι, εντάξει. Υπάρχει κάποιος που βάλει μια πρόταση, δεν έχει κάνει ποτέ κάτι σχετικό πριν, δεν πήρε αρκετούς πόντους, ας το ξεφορτωθούμε και ας δούμε μια πιο τροποποιημένη επιτυχία, ε, μάλλον ε, πρόταση. πολλοί ερευνητές που δεν βλέπουν μέλλον στο εθνικό επίπεδο υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότηση για πώς τα καταφέρουν ευρωπαϊκά. Πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερα χρήματα. Έχαμε κάποιες ακροάσεις με εκπροσώπους από στις διάφορες χώρες. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για το θέμα της οριμότητας του εθνικού συστήματος ε, και άρα δεν μπορούν να διαχειριστούν τις σωστές προτάσεις ή δεν μπορούν να τις συνδέσουν μεταξύ τους ή μπορεί κάποιες έρευνες να είναι καλές σε εθνικό επίπεδο και να ξεμπερδεύει, να τελειώνει. αναλύσαμε τα σχήματα κινητικότητας ε, τα οποία κινούνται βόρειος, ε, δεν ε, πάνε νοτίως. Πολλοί νέοι μελετητές πάνε στη Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία που είναι μεταβατικές χώρες και όλοι πήγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι το σχήμα μετανάστευσης, τώρα με το Brexit ίσως να αλλάξει πρόκειται για αφηγή κεφάλων ή για κυκλική κίνηση. Πρέπει να δούμε και αν ξαναέρχονται πίσω στις χώρες τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό στον τομέα των κινήτρων. Τώρα, μιλήσαμε για επιπτώσεις της συγκέντρωσης των διορθωτικών ταμείων. Ναι, κάποιες φορές έχουμε την εντύπωση ότι οι πολιτικές μπορεί να συγκρούνται μεταξύ τους, ας πούμε τα διορθωτικά ταμεία με βάσει την αρχή της αριστείας, αλλά στην πράξη δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο ως πρόγραμμα για τα διευθυντικά ταμεία. Θα πρέπει να είναι ξεχωριστά. Οι στρατηγικές, οι ευφύς στρατηγικές μπορεί να είναι ένας τρόπος να φύγουμε από αυτό. Γιατί αν υπάρχουν επιπτώσεις συγκέντρωσης, είναι αντιπαραγωγικό αυτό, γιατί ε, δεν έχει περισσότερη εντοχή αυτό το σύστημα. Περισσότερο έχει να κάνει λοιπόν με την ε, με ένα ε, ανθεκτικό εθνικό σύστημα καινοτομία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τις πατρίσεις σας και τώρα έχουμε την κυρία Ζόνεβελτε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ήταν μια ερώτηση σχετική με, το πώς θα πρέπει να οθηθούν τα κράτη-μέλη για επενδύσεις στην έρευνα. Ίσως θα μπορούσε να προσκληθεί ένα κράτος μέλος να προκαταβάλει χρήματα στον ορίζοντα με ένα μόνο σύνολο κανόνων, κανόνων συμμετοχής δηλαδή στο ορίζον, και να προδιατίθεται και πιο γεννόδωρος προπολογισμό. Ίσως αυτό ήταν μια ιδέα. Γιατί έτσι τα κράτη-μέλη θα βλέπουν τα δικά του σχέδια, τα δικά του έργα, πιο στενά συνδεδεμένα με το ορίζον. Γιατί κάποια κράτη έχουν λιγότερα έργα από άλλα. Ένα από τα πράγματα που ανακαλύψαμε σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όταν αρχίσουμε να συζητούμε για το πώς οργανώνουμε τη δουλειά μας στο δικό μας πανεπιστήμιο και άλλοι μας λένε πώς εξασφαλίζουν υποστήριξη κτλ. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για όλους και έτσι μπορεί νομίζω και να επενδύσει ένα πανεπιστήμιο στο κλείσιμο του κενού έρευνας και καινοτομίας. Επίσης καινούρια προγράμματα της Εθνικής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης μαζί βέβαια με άλλες εθνικές υπηρεσίες μπορούν να πάρουν μεγαλύτερη ορατότητα. Χορηγοί μπορούν να έρθουν ε, στη Γάνδη, και να δούνε πώς δουλεύει. το δίδαγμα από την ε, λειτουργία του 7ου προγράμματος πλαισίου ήταν ότι φέρνει αποτελέσματα, έφερε αποτελέσματα, δημιούργησε θέσει εργασία πολλέ, ε, συνέβαλε σημαντικά στην, ε, στο ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να το αλλάξουμε λοιπόν, αφού αναμένεται ότι θα κάνει κάτι καλύτερο, ακόμα το ορίζουν με την εστίαση στην καινοτομία, γιατί να το αλλάξουμε. δάνεια για την κυρία Ρούις που με κάλεσε να δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες για τα δάνεια. Εμείς έχουμε δάνεια μόνο για τους ε, φοιτητές μας και συναφείς δραστηριότητες ή επιχειρήσεις, επομένως χωρίς να είμαστε κατά των δανειών ως πανεπιστήμιο, δεν ευνοούμε τη χρήση του ερευνητικού προϋπολογισμού μόνο και μόνο για να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες για τα δάνεια. Υποστηρίζουμε βεβαίως τις προτάσεις Επιτροπής για το EIC ε και βλέπουμε ότι υπάρχει κενό. Στο επίκεντρο όμως του ορίζον πρέπει να παραμείνει έρευνα μαζί με την καινοτομία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους επιρρογνώμονές μας. για τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια. Και πάμε στο τρίτο θέμα, συνεργατικές σχέσεις, ανάπτυξη δυναμικού, συνοχή ή Ευρώπη δύο ταχυτήτων και θα παρακαλέσω τον κύριο Κρίστοφ να λάβει το λόγο. Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Πολωνία, Φιλανδία, Ενωμένο Βασίλειο. Έχετε πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία από ό,τι βλέπουμε. Και είστε ειδικό επίσης στους τομείς του παρατηρητηρίου της έρευνας και της καινοτομίας. Έχετε αναλάβει εκθέσεις αξιολόγησης ομοτήμων, Φερρυπίνου Πουδαπέστη, και διατελείται διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ο Ευρωπαϊκός λοιπόν τομέας τροφίμων. Που έχει την ευθύνη της δημιουργίας νέων προτάσεων για την καινοτομία στα τρόφιμα. Το Νοέμβριο του 2016 μάλιστα εξελέγεται σε αυτήν την θέση. Πολύ πρόσφατα. Έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω δύο διαφορετικά σενάρια συνεργατικές σχέσεις και Ευρώπη των δύο ταχυτήτων που λίγο πολύ καταγράφηκαν νομίζω και από τους προηγούμενους ομιλητές. Πριν από δύο εβδομάδες μόλις ε, σημειώσαμε μια σημαντική επιτυχία η οποία νομίζω δείχνει τη σημασία των συνεργατικών σχέσεων στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν οι φωτογραφίες που βλέπετε εδώ αυτές που λέμε οικογενειακές φωτογραφίες είναι ίσως τελευταίες που θα έχουμε εδώ βλέπετε τα ευτυχισμένα πρόσωπα των ε, ευεργετηθέντων από τα προγράμματα αυτά που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από πολλές χώρες, από τη Γερμανία, την Ελβατία, την Ισπανία και πολλές άλλες, που με κοινέ προσπάθειες δημιουργήσαν ε, συνεργατικές σχέσεις για, τον, για την έρευνα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα που έχω να σας παρουσιάσω χαράζουν μια κάπως πιο ζωφερή εικόνα. Αν συγκρίνουμε λοιπόν στατιστικές και την κατανομή της χρηματοδότησης και μάλιστα συγκρίνουμε τη χρηματοδότηση του Οριζόντα 2020 με τις πρόσφατες επιδόσεις της έρευνας, Δυστυχώς η υπόθεση ότι υπάρχει ακόμη η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων επιβεβαιώνεται τα μάλα. Είχαμε λοιπόν τις 200 πρώτες προκηρύξεις του ορίζον 2020 με 4,68% μόνο από τις ε, χώρες, ε, τις 13 χώρες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Κάποιες χώρες μας λένε βέβαια έχουν λιγότερο ορίμα συστήματα έρευνας και ευχαριστώ τον κύριο Μαρτινότση, τον καθηγητή για την επισήμανση, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα από το οποίο υποφέρει η έρευνα σε αυτές τις χώρες. Εάν κοιτάξουμε τα χρόνια μεταξύ του 2006 και του 2015, οι χώρες ε, της Ευρώπης, 28 χώρες μέλη, έχουν ε, σημαντικά ενισχύσει την συμμετοχή τους στην χρηματοδότηση και ιδιαίτερα την έρευνα τη χρηματοδότηση της έρευνας. Αν δούμε τις στατιστικές που αφορούν τα πρώτα 15 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μάλλον υψηλότερα τα ποσοστά αυτά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανάλυσης βέβαια των στατιστικών δεδομένων για την απόδοση της καινοτομία. Και έτσι, εάν συγκρίνουμε διαφορετικούς τύπους απόδοσης output δηλαδή της καινοτομία χάρη στο ορίζον 2020 και τα ποσά που χορηγήθηκαν στις διάφορες χώρες. Η υπόθεση, η διαφορά ε, υπεροχή στην έρευνα θα έπρεπε να οδηγεί σε ισότιμα επίπεδα για τις 15 χώρες ε, της Ευρώπης και για τις 13, δηλαδή το μπλε αντίστοιχα και το πορτοκαλί κομμάτι του χάρτη. Αν όμως κοιτάξουμε διαφορετικούς τύπους ερευνητικών δεδομένων, ε, αποκλήσεις καταγράφονται επιστημονικές δημοσιεύσεις για κάθε χίλια ευρώ, για τα χίλια ευρώ που θα πάρει κανείς από τη χρηματοδότηση. Οι 13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις όπως επίσης και οι παραπομπές επιστημονικά ε, πονήματα παρουσιάζουν πολύ θετικότερη εικόνα ε, οι 13 τελευταίες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτές που έχουν πάρει και το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία το ίδιο και για, τις τα εσωτερικά μοντέλα, όπου μόνο η Γερμανία φτάνει σε επίπεδα των 13 νεότερων κρατών μελών. Το ίδιο έχει να κάνει και με τις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι εξισορροπημένη ε, η απόδοση της χρηματοδότησης του ορίζον 2020, όπως δεν είναι και η χρηματοδότηση ισότιμα κατανεμημένη. Αν αυτή γινόταν ε, ε, με βάση την αριστεία, θα ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα. Εδώ σας δείχνουμε πόσο έντονες είναι οι διαφορές. Και εγώ ως Πολωνό... θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το παράδειγμα της Πολωνίας που έχει διπλασιάσει τη χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη τα τελευταία δέκα χρόνια και ιδιαίτερα το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δαπανών για την έρευνα και ανάπτυξη. Ταυτόχρονα. Και ενώ κατέστη δυνατό να αρθούμε στο ύψος των προσδοκιών που είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση και τις προβλέψεις της χρηματοδότησης του Horizon 2020 και είμαστε σε επίπεδο υψηλότερο του 1% ε, λόγου επί του ΑΕΠ σε δαπάνες. Ταυτόχρονα το μερίδιο χρηματοδότησης που έφτασε σε δικαιούχους από την Πολωνία με το πρόγραμμα πλαίσιο 6 και αντίστοιχα το 7 και το Horizon 2020 έχει πέσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξάνονται οι εθνικές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ αντίστροφα ακριβώς καταγράφεται η τάση όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Τρεις λόγοι μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό. Αφενός και ίσως ο καλύτερος τρόπος να το εξηγήσουμε είναι να παραθέσουμε τα λόγια μεγάλου ερευνητή της βιοιατρικής από το Λονδίνο που έλεγε ότι το ορίζον 2020 έχει έναν τρόπο αντιμετώπισης της αμοιβή των ερευνητών από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης είναι και παραθέτω το ακατονόμαστο σύστημα υποαποζημίωσης, υποαμοιβής των ερευνητών από τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Αυτό το παράδειγμα το βλέπουμε ξεκάθαρα στην Πολωνία και στον ορίζοντα 2020 ακόμα περισσότερο βλέπουμε σχεδόν να τιμωρούμαστε εάν έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Ο μισθός είναι ούτως ή άλλως περιορισμένος, αλλά ε, ο ερευνητής μπορεί να πάρει ε, ένα πριν παραπάνω, ένα μπόνους παραπάνω, ώστε να ξεπεράσει τα επίπεδα, όρι, ε, τα επίπεδα των αμοιβών που αναγνωρίζει το σύστημα Horizon 2020. Ένας άλλος λόγος να εξηγήσουμε αυτές τις αποκλήσεις και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα πάλι σχετικό με την Πολωνία ο επικεφαλής μάλιστα του Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου, του κυρίου δηλαδή χρηματοδότη έρευνας και ανάπτυξης, το εξήγησε, ε, μας είπε ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε εθνικά κονδύλια και όχι ε, χορηγίες από το ERC, γιατί είναι πολύ χαμηλότερες αυτές από ό,τι θα μπορούσε ένας ερευνητής να εξασφαλίσει από τα εθνικά από την εθνική χρηματοδότηση της έρευνας. Άρα κάτι πρέπει να πηγαίνει πολύ πολύ στραβά στις διαδικασίες και το σχεδιασμό του ορίζοντα 2020. I think we, we will have a question time in, in, in, in 15 minutes. Okay, okay. Οι ερωτήσει θα έρθουν σε λίγο. Έχουμε, υπάρχουν ασφαλώς διαφορετικοί τρόποι, θα μου πείτε, να ε, εξηγηθούν τα προβλήματα, αλλά αφορούν και, τους, και τα 13 νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει επαρκείς απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την έποψη των ερευνητών των πανεπιστημιακών από τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα είναι απλούστατα οι εργαζόμενοι ερευνητέ, ε, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, θεωρούν ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται, ότι κανεί δεν δίνει σημασία και ότι, εν περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν και συγκεκριμένα συμφέροντα που οδηγούν κάποιους θεσμούς να μην θέλουν να ανοίξει συζήτηση στα θέματα αυτά. με κάποιες συνομιλίες που είχαμε με φίλους μας στο Κοινοβούλιο διαπιστώθηκε ότι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πάπους Πόρα της Ρουμανίας αποφάσισαν να μην υπογράψουν συμφωνία για χορηγία από το Horizon 2020 γιατί ήδη επίστωσαν ότι ο προϋπολογισμός που θα τους χορηγούνταν δεν αρκούσε για να καλύψουν τις προσωπικές δαπάνες με βάση τους μισθούς που στηρίζονται στις επιδόσεις. Πρόβλημα λοιπόν είναι η μισθή, αλλά υπάρχει και άλλο πρόβλημα πιο ουσιαστικό. Φανταστείτε μια τάξη με 15 παιδιά που παίζουν μαζί εδώ και μερικά χρόνια. Και σε αυτήν την τάξη μετά τα 15 παιδιά μπαίνουν άλλα 13 παιδιά. και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε αυτά τα 15 παλαιότερα παιδιά να παίξουν και με τα καινούργια παιδάκια, τα 13. Αλλά κάποια δεν ενδιαφέρονται να παίξουν με αυτά τα καινούργια παιδάκια. Το κύριο πρόβλημα, το κύριο για τα ερευνητικά Ινστιτούτα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ή νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν τα καλούν να παίξουν. Ή δεν ε, λαμβάνουν συστάσεις να γίνουν μέλη συμπράξεων. Το βλέπουμε αυτό και η κυρία Σόνεφελτ μας είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ε, ε, χρηματοδότηση δικτύωσης στο ορίζον 2020, η αρχική υποστήριξη των ε, δραστηριοτήτων. Ναι, μάλλον, μάλλον θα συμφωνήσω. Δεν θέλουμε παραπάνω χρήματα για τα ταξίδια ή προσωπικές δαπάνες, αλλά θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωριστεί και η όποια αριστεία η επιστημονική υπάρχει στις χώρες μας. Συμβάλλουμε και εμείς στις επιστημονικές ε, συμπράξεις. Και αν πάμε εδώ πέρα που βλέπετε τις μπλε γραμμές και τη δικτύωση εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των 15 παλαιότερων κρατών είναι πολύ πυκνό το δίκτυο, ενώ είναι πολύ πιο αραιό μεταξύ των 13 νεωτέρων κρατών. Και αν ιδιαίτερα κοιτάξετε κάποιες μεμονωμένες χώρες, οι ισπανία η Ελλάδα τείνουν να συμμετέχουν σε πολλές από τις συμπράξεις. Βλέπετε αυτές τις λεπτές, λεπτές γραμμούλες που δείχνουν επανειλημμένους δεσμούς μεταξύ κρατών του ορίζοντα 2020, ενώ χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εστονία, η Κροατία απλώς δεν προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις ε, συμπράξεις και να και θα δείτε πίσω σε διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν. Μόνο εννέα έχουν, συγκαταλέγουν μέλη της Ευρώπης ε, των 13 νεωτέρων και μάλιστα κρατικά από αυτά τα κράτη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν τα περισσότερα χρήματα πάρει στην Ευρώπη το 15. Και εν τέλει, αν σκεφτούμε τρόπους αντιμετώπισης ε, των ε, προκλήσεων προς το σχεδιασμό του ορίζοντα 2020, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω τρεις συγκεκριμένε προτάσεις. Αφενός με εναλλακτική ε, νομοθεσία, εναλλακτικούς κανόνες, ώστε να γίνουν αυτές οι διαφορικές βελτιώσεις των ε, μισθών των ερευνητών ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, προαγωγή της συμμετοχής των άξιων ε, εταίρων στις διάφορες συμπράξεις, Φερρυπίν, ε, το παράδειγμα που σας έδωσα θα μπορούσατε να το δείτε σαν κάτι το ισοδυνάμο με την διάκριση για λόγους φίλου Δεν προσκαλούνται στα, στις συμπράξεις για την έρευνα ερευνητές από τα 13 νεότερα κράτη-μέλη. Και βέβαια χρειάζεται και ευελιξία για να καλυφθούν οι... τα κενά αυτά. Καλώς λέω πρόεδρος και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ινακής Αν Σεμπαστιάν. έρευνα καινοτομία εκνάλια. Πρόσφατα, το Μάρτιο του 2016 αναλάβατε, αλλά ήσασταν και βιομηχανικός ερευνητής μηχανολογίας του Πανεπιστήμιου τη Ναβάρα, είχατε ευθύνε για την ε, διοίκηση επιχειρήσεων, Ήσασταν στις Φλατρόνικ για 16 χρόνια και δύο χρόνια από το 8 έως το 10 ήσασταν Technology και Market Manager της Technalia Corporation που δημιούργησε 8 τεχνολογικά κέντρα και διάφορες βέβαια spin-offs επιχειρήσεις. Έχετε συμμετάσχει διάφορες εταιρικέ σχέσεις ως μέλος των ε, διοικητικών συμβουλίων και το καθεξής. Ναι, να το δούμε λοιπόν πώς είναι αυτό το μέσον FP9. Ένα εργαλείο λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ε, a, Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μας δώσατε την ευκαιρία όχι σε μένα, όχι στην τεκνάλια ε, και όχι μόνο σε μένα. Μιλώ στο όνομα των 350 κέντρων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τεχνολογικών Κέντρων RTOs. Οπότε μιλώ στο όνομα της RTO, της ARTO, ΕΑΡΤΟ, συγγνώμη. Δύο λόγια για την Τεκνάλια, που είναι μια οργάνωση εφαρμοσμένης έρευνας που έχει σκοπό να μετατρέψει την τεχνολογία σε ΑΕΠ και Βεβαίω ε, εδώ συναντούμε τεχνολογία όλων των ε, μελών της ΕΑΡΤΟ, πάνω από 105.000 ερευνητές, 350 κέντρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αφιερώνουν το ταλέντο τους, την προσπάθειά τους καθημερινά έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι πιο ανταγωνιστική. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και σε κάποια ερωτήματα που έγιναν προηγουμένως για το ποια, πρέπει να είναι η αποστολή, ο σκοπός του προγράμματος πλαισίου. Εμείς πιστεύουμε ότι το, το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Διότι είναι δύσκολο να αποσυνδέσουμε τη δυνατότητα του να ανταγωνιστεί κάποιος με το να έχει ε, ε ποιότητα ζωής ε, με το να έχουμε μια κοινωνία δηλαδή που να είναι η καλύτερη για να ζήσει κάποιος. Το πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν είναι ε, η λιδία λίθος ε, του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Οικοδόμησης. Το πρόγραμμα πλαίσιο, επαναλαμβάνω, είναι η λιδία λίθος ε, της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, διότι η Ευρώπη εφόσον εξετάσει κανεί τα στοιχεία, δεν παράγει καινοτομία ή όχι τόσο όσο οι υπόλοιποι. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως περιφέρεια. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος ο Επίτροπος. Που α, μιλώντας για τις διαφορές μεταξύ του ορίζοντα 2020 και του FP7 ε, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη αύξηση του προπολογισμού πήγε προς την αριστεία και την έρευνα. Εγώ δεν νομίζω ότι η βασική έρευνα έχασε. Εδώ φτιάξαμε πυλώνες πιο ισορροπημένους, αλλά εκεί όπου έχουμε μεγαλύτερες προκλήσεις είναι εκεί όπου προσπαθούμε η καινοτομία να φτάσει έως την αγορά. Είμαστε λοιπόν σε αυτούς τους καταλόγους που καθορίζουν ε, οι επιχειρήσεις ε, και οι προσπάθειες που δημιουργούν πλούτο και δημιουργούν ε, και απασχόληση. Ορισμένες φορές δημιουργούμε απασχόληση, δημιουργούμε ε, πλούτο και ανάπτυξη, αλλά ξεχνάμε, τα άτομα, τους ανθρώπους. Αλλά όταν δημιουργούμε θέσει απασχόληση, δεν ξεχνάμε του ε, ανθρώπου, του θυμόμαστε. Εγώ έρχομαι από την Ισπανία και κάτι ξέρουμε εμεί από τι, σημαίνει ανεργία σε τέτοια υψηλά ποσοστά. Εδώ βλέπετε το κατάλογο της MIT, η πρώτη, ελληνική, η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία είναι 28η. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποιος είναι ο σκοπός της καινοτομίας και πραγματικά θεωρούμε ότι η θα πρεπει λοιπον να σκεφτουμε ποιο ειναι ο σκοπος της καινοτομια και πραγματικα θεωρουμε οτι η καινοτομια θα πρέπει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να βοηθήσει στην επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και ε, αυτό είναι που θα κάνει την ευρωπαϊκή κοινωνία την καλύτερη του κόσμου. Για μας εδώ υπάρχει μια ζυγαριά που είναι πολύ σημαντική. Εγώ εδώ εκπροσωπώ τους τα, τα ευρωπαϊκά, τα, τα, τα κέντρα, τα e, e τους RTOs. Παίζουμε ένα ρόλο κλειδί λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτές τις αλυσίδες αξίας. Είμαστε συνδεδεμένοι και με τους ερευνητέ και ε, με τις επιχειρήσεις και με τους πολιτικούς θύνοντες. Έχουμε τρεις ε, σκοπούς. Είμαστε εξαιρετικά ενεργοί στον τομέα της έντονας και ανάπτυξης. Δοκιμάζουμε λύσεις απέναντι στις κοινωνικές προκλήσεις και υποστηρίζουμε και την ε, βιομηχανία για να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική. Είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος από τον TRL3 προς την trl από την επιστήμη προς την καινοτομία στην αγορά. Θέλουμε να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε την επιστήμη και την έρευνα πιο κοντά στην αγορά. Το σημείο κλειδί για την καινοτομία, ο παράγοντα κλειδί είναι η επιχείρηση. Εμεί είμαστε συνδεμένοι με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα. Όταν ένα μέλος της ΕΑΡΤΟ συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο project του ορίζοντα 2020, το ποσοστό των επιχειρήσεων είναι 6% πάνω από το μέσο όρο. Η δυνατότητα λοιπόν να παρασύρουμε μαζί μας ε, επιχειρήσεις στα προγράμματα αυτά, που πρέπει να είναι και στόχος του προγράμματος πλαισίου, αυτή η δυνατότητα είναι πολύ πιο μεγάλη όταν υπάρχουν τα, αυτά τα τεχνολογικά κέντρα. Πιστεύω πραγματικά ότι τα κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ε, ενεργούς παράγοντες ε, σε τεφάσεις προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Συμμετέχουμε ανελιπώς σε μια σειρά από εργασίες στον πολιτικό, περιφερειακό, τοπικό, εθνικό τομέα, αλλά επίπεδο, μάλλον και σε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική έρευνα και ανάπτυξη. Είμαστε συνδεδεμένοι και με τι επιχειρήσει. Γνωρίζουμε ποια είναι, είναι τα προβλήματά του, ποιε είναι οι προκλήσει που έχουν να αντιμετωπίσουν, τα προβλήματα ανταγωνιστικότητα που αντιμετωπίζουν. Και βεβαίω είμαστε, είμαστε παρόντε και στα διάφορα μέσα, στα διάφορα εργαλεία τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ευρωπαϊκέ πλατφόρμες. Δηλαδή είμαστε έτσι ένα, ε, ένα συνδετικός κρίκος και μπορούμε να συνεισφέρουμε σημαντικά για να καθοριστούν προτεραιότητες στον τομέα έρευνα και ανάπτυξης. Θα ήθελα τα τελευταία λεπτά της παρουσίασής μου να κάνω κάποιες συστάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο. Εδώ ε, υπάρχει η εμπειρία ετών συμμετοχής στα προγράμματα πλαίσιο κατά κάποιο τρόπο αυτή την εμπειρία την έχουμε εδώ μεταφράσει σε συστάσεις. Καταρχήν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον αντίκτυπο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να δημιουργήσουμε σαφή ωφέλη για την κοινωνία. Η, επιστημονική κοινότητα, η κοινότητα των ερευνητών πρέπει να συνάψει ένα νέο συμβόλαιο με την κοινωνία και να δεσμευτεί για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι απαραίτητο. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε μέσω τη οικονομική ανάπτυξη, μέσω τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και μέσω τη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μα. Δεύτερον, εμείς είμαστε υπέρ μιας συνεργατικής προσέγγισης, μοντέλα δηλαδή που ενισχύουν τη συνεργασία. Είναι άλλο ένα μάθημα από την ιστορία των διαφόρων προγραμμάτων πλαίσιο. Εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Ναι, δεν έχω τελειώσει, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα καινοτομία τη Ευρώπη. Οι υποδομές καινοτομία που έχουμε, τα διάφορα εργαλεία, πιστεύουμε ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο καταλήτη αυτό το πρόγραμμα στην Ευρώπη. Μπορούμε εδώ να συνδυάσουμε τα διάφορα εργαλεία, τα διάφορα μέσα έτσι ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η δυνατότητα καινοτομία. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών του κλάδου που εξασφαλίζει την καινοτομία. Τώρα, σε σχέση με το δίλημα στο οποίο έγινε αναφορά προηγουμένω μεταξύ ε, χορηγιών, υποτροφιών, τους πάντων ενισχύσεων και δανείων, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις υποτροφίες, της ενισχύσεις. Στην Ισπανία είχαμε μια μετάβαση τα τελευταία χρόνια από τη χρηματοδότηση προ τα δάνεια και ε, απέτυχε. Σε γενικές γραμμέ απέτυχε. Υπάρχει εδώ μια ολόκληρη γραμμή η οποία δεν έχει τελεστεί και πρόκειται για μια στρατηγική επιστροφή τώρα στην χρηματοδότηση διότι δεν δίνονται υπαρκή κίνητρα για να λάβει χώρα δανειοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε μια καλή χρήση των υποδομών που έχουμε στη διάθεσή μας, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ μπορεί να είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Τέλος, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες απλοποίησης που έχουν ξεκινήσει στα πλαίσια του 2020. Και κάτι τελευταίο. να πω κάτι για το ποσοστό επιτυχίας. Τέσσερα αριθμητικά στοιχεία έως τώρα είχαμε 109.000 προτάσεις ε, στο πλαίσιο του 2020. 13.000 ε, ε, χρηματοδοτήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι 95.000 δεν χρηματοδοτήθηκαν. 50 εκατομμύρια ώρες εργασίας, έτσι. 30.000 ερευνητές χρειαζόμαστε για να μπορέσουν να υποβάλουν αυτές τις προτάσεις. Μιλάμε για ένα κόστος των 5 δις ευρώ. Πρέπει να προσθέσουμε, προσθέσουμε βεβαίως και το τι θα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν έκαναν αυτό. Και αυτό είναι απώλεια. Λοιπόν, μιλάμε για την επιτυχία των καλών προγραμμάτων. Τα μισά από τα προγράμματα αυτά η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πολύ καλά. Θα πρέπει λοιπόν πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το θέμα της αριστείας. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι όλη αυτή η επένδυση που έχει γίνει δεν μπορούμε τώρα να την καταστρέψουμε και να τη χάσουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Η κυρία Καπεθόν Ρουίς, η κυρία, μας, η κυρία εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ τους μιλητές και σύντομα θα μιλήσω γιατί φαντάζομαι όλοι θα θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Στον κύριο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας της Πολωνίας νομίζω πως έθεσε επιτάπητος ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα το οποίο συζητάμε και που είναι προφανές και έχει μάλλον υποδεχτεί και με βάση την τελευταία μας αποστολή στην Ισπανία και στην Πορτοχαλία και τέθη το ζήτημα είναι το θέμα ακριβώς της συνοχής. Δηλαδή όταν μιλάμε για δύο ταχύτητες ε, και Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε, να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο που έχουν τα προγραμματά μας, τον αντίκτυπο για την αντιγωνιστικότητα, αλλά και στη συνοχή. Είναι αλήθεια ότι το ποσοστό συμμετοχής κάπως έχει βελτιωθεί στις χώρες που σιγά σιγά μπαίνουν στο πρόγραμμα, αλλά είναι πιθανό να μην επαρκεί και θα πρέπει εξ αρχής να, να θεωρήσουμε ότι είναι αυτό αυτονόητο ότι οποιοδήποτε θέλει σε εθνικό επίπεδο μπορεί να ενταχθεί. Θα πρέπει λοιπόν να μην ε, δημιουργηθεί μια ελληματική δομή όπως προς αυτή την, την έννοια. Έπειτα εστιάζουμε και συγκεντρώνουμε την αριστεία και έχουμε φτιάξει κάποιες περιοχές αριστείες. Θα μπορούσαμε να βαθύνουμε σε αυτό. η ερευνητική δομή σε εθνικό επίπεδο πιστεύω ότι πρέπει να βαθενθεί ή η ίδια η δομή ε, και η διάρθρωση του προγράμματος ορίζοντος 2020 ε, κατά, με βάση το κατά πόσο θέλουμε ή όχι να αποκλείει. Και μετά κάνατε λόγο για φυγή εγκεφάλων. Φυγή εγκεφάλων όταν μιλάμε λέμε ε, συνήθως ότι πρόκειται για φυγή εγκεφάλων εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πρέπει να προσεγγίσουμε και την Στη κινητικότητα εντό του ευρωπαϊκού χώρου. Τη δυνατότητα που έχουν οι επιστήμονε να μετακινούνται από μια χώρα στην άλλη, ε, α πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία, πώ μπορούμε να δώσουμε κίνητρο στι ερευνητέ που προετοιμάζονται σε αυτέ τι χώρε και που προσπαθούν να συμμετέχουν σε πιο σημαντικά προγράμματα μέσα στον ορίζοντα 2020 να μην μετακινηθούν από τη μια χώρα και φύγουν τελικά και τελικά το κριτήριο να είναι μόνο το οικονομικό κριτήριο. Πιστεύω πως αυτό το θέμα πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα, για τον εισηγητή του Στεκνάλια και από πλευρά τη ΕΑΡΤΟ, εσεί αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα για το κατά πόσο θεωρούμε ισορροπημένου του πυλώνε. Το κομμάτι του πρώτου πυλώνα, της αριστείας, ε, της ε, βασικής έρευνας θα πρέπει να καλύπτεται. Εγώ από αυτή την άποψη αυτό που θέλω να πω είναι να δώσω ένα μήνυμα που είναι η γνώμη μου. Πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την ανάγκη διατήρησης των πυλώνων ε, του δεύτερου και του τρίτου. Είναι αυτό θεμητό και σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον πρώτο πυλώνα να αποδυναμωθεί. Θα πρέπει δηλαδή να διερωτηθούμε εάν και μήπως ε, βαρύνουμε το ένα μέσο εις βάρος του άλλου, ε, μάλλον υπέρ του άλλου. Νομίζω λοιπόν πως η βασική γνώση είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και να παραμείνει και να προσπαθήσουμε να τον ισχύσουμε την επιστημονική σκέψη, να υπάρξει δηλαδή Έχουμε πολύ καλή βασική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε πρόβλημα γιατί η βιομηχανία δεν μπορεί να μετατρέψει αυτές τις γνώσεις σε πραγματική εμ, να υλοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, να τη μετατρέψει σε, σε εφαρμοσμένη έρευνα, ε, σε κάτι το πρακτικό. Έχω λοιπόν συγκεκριμένε ερωτήσει. Όταν λέτε ότι ο αντίκτυπο ε, ο τεχνολογικό ε, για την πρόθεση της καινοτομία μέσα στη βιομηχανία. Όταν μιλάτε εσείς για αντίκτυπο, τι λέτε προς ε, εγκύτητα περιφερειακή, εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις ή πώς ε, μεταφέρεται η γνώση ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία. Για ποια βιομηχανία μιλάτε, για ποιο μάλλον αντίκτυπο μιλάτε. Έπειτα για τη σημασία του σήματος αριστείας, αλλά τι είδου ε, αξιολόγηση θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ εξαντλητική προσέγγιση του, α, της εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να το αναλύσουμε και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε σύστημα αξιολόγησης ε, ώστε να μπορούμε να ζητήσουμε πιο σημαντική ανάπτυξη το project για να μπορέσουμε όντως να κατευθύνουμε χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό εκεί όπου χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σελέρ πριν από μερικά χρόνια εισηγητής του Ορίζον 2020. Έχετε το λόγο. Συνήθω δεν κάνω σχόλια. Αλλά μια και ο καθηγητής από τη Βαρσοβία είπε ότι είπε αυτά που είπε και επειδή παρακολουθώ τη συζήτηση εδώ και 5-10 χρόνια. Η η εικόνα που μας παρουσιάζεται για τα 13 νότερα κράτη δεν είναι μια μόνιμη εικόνα, δεν είναι συνεπής ότι δεν έχουν το 3% του κοινού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητες έρευνα και ανάπτυξη. Οφείλεται στο ότι έχουν μειωθεί οι δραστηριότητες έρευνα και ανάπτυξη για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 1%. με ένα σταθερό ποσοστό 0,4-0,6%. Λοιπόν, το τι σχέση έχει η συμμετοχή στο 2020 είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Εμείς αρχικά είχαμε προτείνει από το Κοινοβούλιο για τα κράτη-μέλη και δεν θέλω να ξανανοίξω αυτή τη συζήτηση γιατί από κοιτού κοινού έχει γίνει αυτή η συζήτηση η διεύρυνση της συμμετοχής να μην κρίνεται με στατιστικού όρους. Είναι λογικό να γίνεται η διεύρυνση πιο πολύ ε, στα παλαιότερα κράτη-μέλη, διότι οι φυστάμενα όργανα και θεσμοί των παλαιότερων κρατών μελών ιδρύουν νέε σχέσεις ε, για να έχουν τη δικτύωση με τα νεότερα. Έτσι λοιπόν εξηγείται και με τα προγράμματα αδελφοποίησης και τα λοιπά το ίδιο πράγμα είναι. Πολλαπλασιάζουν όπως εκ τούτου τα παλαιότερα ε, κράτη και ερευνητικά κέντρα κρατών ε, τις διασυνδέσεις τους. Είχαμε λοιπόν, πρέπει να σας πω, τεράστια αντίσταση και δει από την Πολωνία γιατί θέλει να κρατήσει τα πάντα στα διαρθρωτικά ταμεία. Είχαμε καυγάδες εδώ μέσα, πολύ σκληρούς αγώνες των 13 νεωτέρων κρατών γιατί λέγανε ότι ένα νέο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ε, θα ήταν πιο δύσκολο ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία ήταν εύκολο να κατανεμηθούν. Ε, στα κράτη-μέλη. Παρακολούθησα τα στοιχεία σας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε διαφοροποίηση μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας καταρχάς. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ε, τα νεότερα κράτη-μέλη με χαμηλότερη βιομηχανική βάση, με πιο ασθενή βιομηχανική βάση, δεν μπορούν να προσελκύσουν πολλά χρήματα από το ορίζον 2020 γιατί υπάρχει ένα περιθώριο παρέμβασης, ε, μάλλον συμμετοχής των μεγαλύτερων ε, ομίλων, και αεροναυπηγικής κτλ. Αλλά παρακαλώ, ε, μην αρχίσετε να κάνετε απλώ μια έκκληση και να λέτε Α, είναι δυσανάλογα κτλ. Περιμένουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. 10-15 χρόνια περιμένουμε ένα διαρθρωμένο διάλογο και πρόταση συγκεκριμένη τι να κάνουμε. Όλοι μαζί είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα ε, αυτούς τους ψευδείς υπενιγμούς που δεν δίνουν καμία λύση. Βλέπουμε ότι σε πολλές από τις χώρες επικρατούν ακόμη στα ελληνιστικά πανεπιστημιακά πρότυπα και βεβαίως ε, δεν θα δώσουμε μόνο για τους μισθούς ε, χρήματα αλλά για την έρευνα. Γι' αυτό καλό θα να ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα πρέπει τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων να τα αξιοποιήσουμε για να ξεπεράσουμε το πεπαλαιωμένο πανεπιστημιακό σύστημα σε σχέση με το, την ουσιαστική δαπάνη. Και επιμένω γιατί η Πολωνία είχε τεράστια επιτυχία στην αποδιόρθρωση του παλαιού συστήματος των πανεπιστημιακών κέντρων και βλέπουμε ότι όταν μπόρεσαν να απαλλαγούν από τα παλαιά συστήματα, όλα τα κράτη είχαν πολύ καλή επιτυχία. Όταν προσπάθησαν να διατηρήσουν τα παλαιά συστήματα, απέτυχαν. Και αυτό θα εγκαταλείψουμε αυτή την ε, φρασιολογία. Τα κράτη της Βαλτικής, σε παραδείγμα, έχουν εθνικό πρόγραμμα για την δικτύωση εθνικό πρόγραμμα για να ενισχύσουν την παρουσία τους και να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στο ορίζον 2020. Αλλά κράτη-μέλη δεν έχουν. Αυτό λοιπόν έχει άμεσο συσχετισμό με το εάν κανείς έχει μπει σε ένα δίκτυο ή όχι. Δεν υπάρχουν 13 ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κάποιοι από τα, παλαιότερα, από τα 15 παλαιότερα κράτη-μέλη να μπορούσαν λόγω των εθνωτικών ταμείων να ανήκουν μάλλον στα 13 νεότερα, ενώ κάποιοι από τα 13 νεότερα θα δίναν εικόνα των 15 παλαιότερων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βασικό είναι ότι θέλουμε με το σύστημα αυτό να βελτιώσουμε την ποιότητα της ε, δαπάνης έρευνας και τεχνολογίας των ερθωτικών ταμείων. Είναι κάτι το οποίο πολλοί συνάδελφοι εδώ πολέμησαν όταν είπαμε θέλουμε η καινοτομία, η έρευνα να μην χρηματοδοτούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Το ορίζον 2020 τα ερευνητικά ταμεία δεν αληθεύει ότι δεν δίνουν χρήματα στην ε, διαχείριση ε, υπεροχής, παραδείγματι. Υπάρχουν όμως προγράμματα, πρέπει να καταγραφούν προγράμματα και το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο τι είπανε τα 13 νεότερα κράτη. Α, όχι, εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε μόνο το σύστημα ε, των πωλήσεων μόνο να ερευνηθεί πρόταση από το Συμβούλιο, από τα εν λόγω 13 κράτη. Δεν είδαμε πουθενά, ρωτήστε και τον κύριο Γκέβιν. Καταλαβαίνουμε τι θέλετε, θέλετε να προχωρήσει το θέμα αυτό. Είναι κάτι που βλέπουμε να ρίχνει τη σκιά του στο πρόγραμμα πλαίσιο 9, αλλά αν αυτό το λέτε ως κατηγορία ότι δεν ε, έχουμε αφήσει να απεοδεσμευτεί το πρόγραμμα, ε, φτάνει πια 15 χρόνια πήρε τις ίδιες κατηγορίες ακόμα. Ευχαριστώ και για συγκεκριμένου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, το, το πράγμα, ε, ε, ναι, ναι, όντως. Δεν θέλω να πω ότι τα 13 νέα κράτη-μέλη δεν ε, φαίνεται να κατορθώνουν να αντιληφθούν γιατί δεν τα προσκαλούν στην προαγωγή της έρευνας. τα παλαιότερα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία ζητούν περισσότερους ερευνητές και ισχυρούς εταίρους. Επομένως το widening participation όπως ένα από τα προγράμματα. Δεν έχει φέρει 100% τα ε, αναμενόμενα αποτελέσματα. Και ίσως αξίζει τον κόπο να κοιτάξουμε προγράμματα όπως το ΕΡΑ, προγράμματα αδελφοποίησης και άλλα. Και να δούμε πώς χρειάζεται τελικά να τροποποιηθούν. προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των νέων κρατών μελών. Και το πρόβλημα για μένα είναι διαφορετικό οι νέοι ερευνητές, όχι μόνο από τα παλαια κρατημέλη, αλλά και την Ισπανία και την Πορτογαλία, Φερρυπίνη, Ανδαλουσία που επισκεφθήκαμε, δυσκολεύονται να αντλήσουν τις επιχορηγήσεις, την αξιολόγηση των ε, έργων, επί που θα πρέπει να επανεξεταστούν. Και εδώ, κύριε, μας έχει ένα ζήτημα πολύ συχνά όταν ε, κατακυρώνεται σε ένα νέο ερευνητή έργο, μπορεί να προκύψει σαν χιονοστιβάδα, επιδότη, επιχορήγηση και για το ερευνητικό έργο και για άλλα πράγματα. Έτσι μια χιονοστιβάδα η οποία θα έπρεπε να εξυπηρετεί την ε, ε, επιβίωση την, ε, τα προστοζήν του νέου ερευνητή. Μια άλλη πτυχή που νομίζω σχετίζεται με τα όσα είπε ο συνάδελφος μπορούσαμε ίσως να κοιτάξουμε, να ενθαρρύνουμε τα κέντρα αριστείας να μετακινηθούν σε δομές των νεότερων κρατών μελών, παραδείγματι. Και έτσι μπορούν και οι άριστοι ερευνητέ να διευκολυνθούν στη συμμετοχή, στη συνεργασία σε ε, έργα τα οποία ωφελούνται από το νέο Συλλογή, Συνοχή, τα Διαρθρωτικό Ταμείο κτλ. Ε, πάντα ε, από τη σκοπιά των 13 νεότερων κρατών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος Μάραγαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα ε, της Ευρώπης των 15, της Ευρώπης των 13 ε, και αυτή η αντίθεση είναι αρκετά αποκαλυπτική, έτσι. Ε, έχει ένα θεαματικό χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ πιο περίπλοκο, είναι πολύ πιο μεγάλες αντιφάσεις τελικά. Δεν θέλω να διαφωνήσω με κάτι, θέλω να προσθέσω κάτι. Υπάρχει ένα πρόβλημα ισορροπία στο ιστορικό της κάθε χώρας. Υπάρχουν επιτυχίες ε, υπάρχουν και δυσκολίες στην ίδια χώρα. Ένα από τα, ναι, μια από τις επιπτώσεις του 2020 είναι ότι επικεντρώνει μεγάλα project ε, σε μεγάλα κέντρα ε, τα οποία όπου υπάρχουν συμπράξεις και αυτό βεβαίως δίνει προτεραιότητε σε κάποια εδάφη, σε κάποιε περιοχέ. Ε, τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία έχει μειωθεί κατά 30% ο προπολογισμό εθνικό για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην 2020 είναι πολύ πιο υψηλό το ποσοστό. Αυτό που οδηγεί λοιπόν, ε, ο το 2020 πάει εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητε, όπω στην Τεκνάλια. Φυσικά συγχαρητήρια. Ε, με βάση το στόχο το 2020 καινοτομία, βιομηχανία κτλ. Ε, λογικό είναι. Αλλά αυτό, αυτό δημιουργεί ένα κενό, δημιουργεί ένα χάσμα. Στον, στα μικρά project, στο, στη βασική έρευνα, στον πανεπιστημιακό κόσμο. Η ισορροπία μεταξύ των πυλώνων πρέπει να το προστατεύσουμε, όχι αντικαστώντα το πυλώνα 1 από το πυλώνα 2 ή να αλλάξουμε τη βασική έρευνα και να την να την εγκαταστήσουμε από την εφαρμοσμένη. Όχι, πρέπει να προσθέσουμε πράγματα, όχι να αντικαταστήσουμε πράγματα. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδου επιλογέ, να βγάλουμε το ένα, να βάλουμε το άλλο. Και για τον τρίτο πυλώνα τι κοινωνικέ αλλαγέ, ε, αυτό πρέπει να είναι οριζόντιο. Δεν είναι ανεξάρτητο, είναι οριζόντιο. Πρέπει να αφορά όλου του άλλου πυλώνε. Οι πολιτικέ και κοινωνικέ προτεραιότητε πρέπει να αποτελούν ε, κριτήριο για όλου του πυλώνε για τα διάφορα που υπόθηκαν πριν ε, που δείχνουν ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά. Ε, στις πολιτείες αυτό έχει γίνει, έτσι. Έχει εφαρμοστεί αυτή η τακτική και στην τομέα της αριστείας και της κανοτομίας υπάρχει μια συγκέντρωση κάπου σε κάποια σημεία και κατά τα άλλα έρημος. Έτσι, έχει κάποια καταπληκτικά εδάφη οι με τεράστιες δυνατότητες και γύρω-γύρω έρημος δεν νομίζω να πρέπει να είναι αυτός ο στόχος μας για την Ευρώπη. Και ένα άλλο παράδειγμα από την Ισπανία. Μέρος της επιτυχίας ε, του του 2020 στη Γαλλία παραδείγματος χάρη για λόγους ε, ε, υπάρχουν μεγάλα κέντρα που προτιμούν να μην συμμετάσχουν στην όσο 2020. Ή πάνε λιγότερο από ό,τι θα μπορούσαν. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο έρχεται να νοθεύσει κάπως την αξιολόγηση. Και τέλος. Όταν μιλάμε για δάνεια, ε, δάνεια σημαίνει επιστροφή μετά, σημαίνει απόδοση. Εγώ είμαι υπέρ των υποτροφιών, αλλά οι υποτροφίε σημαίνουν, σημαίνουν και, αυτέ, και αυτές αυστηρότητα. Ε, να μπορούμε να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε πού πάνε αυτές οι υποτροφίες και να πιάνουν τόπο. Μάλιστα, η κυρία Βιέρνιγκ έχει το λόγο και οι συγκρίσει των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Κβίντσεβιτς. Κάποια στιγμή μας είπατε ότι τα επιπλέον κονδύλια ε, για τη δικτύωση αλλά και άλλα επιπλέον κονδύλια. Είπατε ότι συμφωνείτε με την κυρία Ζόνεφελντ το προπολογισμό, αλλά παράλληλα μας είπατε ότι η υπηρεσία σας ε, ε, ε, δεν τους αφορά τόσο το θέμα αυτό της δικτύωσης. Πώς σκοπεύετε να το επιλύσετε το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, η κυρία Νίμπλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτηση της συναδέλφου είναι πολύ σωστή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε αυτό. Ότι θα ήταν καλό να μας προτείνουν οι ομιλητές μας πώς βλέπουν τη λύση του προβλήματος. Όχι μόνο να γύρουν ζητήματα μισθών, αλλά και προτάσεις. Και επίσης, Έχετε κανένα θετικό παράδειγμα για τα 13, από τα 13 νεότερα κράτη-μέλη. Έχετε κάποιο να προτείνετε για να δούμε τι πάει καλά και τι στραβά. Γιατί μόνο παράπονα ακούω. Όλα εδώ είναι χάλια ή τα παλαιότερα 15 κράτη-μέλη επωφελούνται. Δεν είχα εγώ τέτοια εντύπωση μέχρι τώρα από άλλα προγράμματα. Έχετε κανένα θετικό παράδειγμα να μας παρουσιάσετε τι έχει πάει καλά, τι έχει φέρει αποτελέσματα στα 13 ε, νεότερα κράτη που θα μπορούσε ως εκ τούτου και να ε, αξιοποιηθεί περισσότερο. Ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο συνάδελφο που είπε ότι θέλει κάποια success story, ας πούμε, ε, από κάποια από τις χώρες που ε, προσχώρησαν το 2004. Υπάρχει ένα σχέδιο στο Βουκαρέστι, εξαιρετικά επιτυχημένο, ένα project, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, στο Βουκουρέστι. Παρεμφερές με το ΣΕΡΝ. Για πρώτη φορά μπορούμε να κάνουμε ε, πειράματα σε ένα τόσο σημαντικό κέντρο αριστείας στην Ανατολική Ευρώπη. Και δεν συμμετέχουν μόνο Ρουμάνοι ερευνητέ σε αυτό, αλλά και από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Πιστεύετε ότι είναι φυσιολογικό ένα ερευνητή ε, από τη Ρουμανία να πληρώνεται 3 ευρώ την ώρα και κάποιο που έρχεται από τη Γερμανία να κερδίζει 50 φορέ περισσότερα ενώ κάνουν την ίδια δουλειά. Θεωρείτε ότι αυτό το, το, το περίφημο παράδειγμα του ταξιτζή, ξέρετε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, αμέσως μετά την επανένωση, ένας ταξιδιώτης έρχονταν από την Ανατολική Γερμανία, πληρώνονταν πέντε φορές λιγότερο από αυτόν που έμενε στη Δυτική. Ενώ και οι δύο εργαζόταν στο Βερολίνο, έκαναν την ίδια δουλειά. Λοιπόν, πρέπει να απομακρυνθούμε από το μοντέλο αυτό και αν θέλουμε να στεφθεί από επιτυχία η συνεργασία, θα πρέπει αυτή η κοινότητα που δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν είναι τόσοι πολλοί ερευνητέ, η κυρία Καπεθόντου είπε κάτι προηγουμένω. Τι ζητάει αυτή η κοινότητα. Ζητάει, σεβασμό και ζητάει την δυνατότητα να εργαστεί. Και να σας πω ότι η ιστορία θα μας δικαιώσει. Διότι οι ερευνητές και οι Ρουμάνοι ερευνητές έχουν συμμετάσχει στην έρευνα στην Ευρώπη. Η Ινσουλίνη αλλά και οι κινητήρες έχουν ε, ανακαλυφθεί από Ρουμάνους και όλα τα αεροπλάνα τα οποία κυκλοφορούν στον ουρανό σήμερα ε, κυκλοφορούν χάρη σε τους κινητήρες που ένας Ρουμάνος. Γι' αυτό πετάνε. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στο θέμα αυτό. Αν θέλουμε ε, να έχουμε επιτυχίες πρέπει να έχουν όλοι ίση μεταχείριση. Έτσι ώστε όλοι να υποφελθούν από αυτά τα ταμεία. Και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σοφοί. Θα πρέπει αυτή η οδηγία να καταργηθεί. Ήρθε ο επίτροπο στο, Βουκα... Βουκουρέστι πριν από ένα μήνα και κατάλαβε ποιε είναι οι δυσκολίες λόγω τη απόφαση αυτή που έχει δημιουργήσει διαφορέ ε, αμοιβή. Ποια, ποια, ποια έρευνα μιλάμε όταν κάποιο λαμβάνει 3 ευρώ την ώρα, πληρώνεται 3 ευρώ την ώρα. Θα πρέπει λοιπόν να παρθούν μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση, διότι τα μέλη των, των πρώην 13, των 13, χωρών της Ένωσης είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριος Κόχλης, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κύριος Έλερ, καλό θα ήταν να ρίξει μια ματιά στην Ευρώπη και να μην κοιτάει μόνο τη Γερμανία. Γιατί εσείς κύριε Έλερ, Κάνατε ερωτήσεις και ζητήσατε αποτελέσματα. Μισθούς, έδρες διεθνών επιχειρήσεων, εφαρμοσμένη έρευνα. κάνατε λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις, δεν θα ξανθυνεζόσασταν τόσο. Θα είχατε μια πολύ καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας. Δεν είναι εύχερης ε, ο υπολογισμός, η αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας των έργων. Εγώ θυμάμαι να εξασφαλίζω τη χρηματοδότηση ενός αρκετά περίτεχνου κλιβάνου ή αλουργίας ε, που όμως τελικά δεν μπόρεσε να ευοδοθεί γιατί ήταν περίπλοκο το σχέδιο και χρειάστηκε εμείς να το πληρώσουμε η μισθοί μας για την ίδια δουλειά και συγκρίνω μεταξύ ε, ε, Τσεχικής Δημοκρατίας και Γερμανίας έχουν σχέση ένα προς τρία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν καλά την ε, πραγματικότητα και μετά ας εξανιστάμεθα. γιατί τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά θέλω να αντιληφθεί κανείς που εδρεύουν αυτές οι επιχειρήσεις. Εγώ είμαι η αλουργός. Έχουμε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ξέρουμε ότι την έρευνα την έχουν στο Βέλγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στις χώρες μας παράγεται το κέρδος. Την Πολωνία, τη Σλοβακία, εν μέρη και τη Γερμανία. Όχι, μιλάω μόνο για την ιαλουργία. Μπορεί η κατάσταση σε άλλους τομείς να είναι διαφορετική. Η εφαρμοσμένη έρευνα στην Ιταλία, Φερρυπίν, μπορεί να ε, είναι πιο δεδομένη στο βορρά και να απουσιάζει πλήρω από τον νότο της χώρας. Υπάρχουν πάντα αποκλήσεις. Και κάτι ακόμη, ένας άνθρωπος μιλούσε και επιτυχή έργα. η τσεχική δημοκρατία είναι υπερδύναμη στα υπερελαφρά αεροσκάφη. Ηλεκτρικό αεροσκάφος επίσης, μια τεράστια επιτυχία, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να παραλυφθεί. Για τον κύριο Έλερ επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ε, απασχολησιμότητας ε, στο ημελουργία είναι αυτό της Γερμανίας, 50.000 εργαζόμενοι στη Γερμανία, 25.000 στην Τσεχία. Η εφαρμοσμένη έρευνα που λαμβάνει χώρα α, στη Γερμανία, αυτό θα σας απαντήσω. Εφαρμοσμένη έρευνα στην ιαλουργία, στην Τσεχική Δημοκρατία δεν υπάρχει. Αλλά εργάτες έχουμε, εργάτες της ιαλουργίας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά λοιπόν μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών. Αυτή η διαφορά από την οποία θέλουμε και να απαλλαγούμε. Θέλουμε να αλλάξουμε, να αντιστρέψουμε την, ε, τις αποκλήσεις στους μισθούς. Με, ακόμα και με τις αυξήσεις που έχουν δώσει στην τσεχική δημοκρατία για τους ερευνητές ε, και επιστήμονες, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν για τη Γερμανία και την Αυστρία που έχουν καλύτερου μισθού. Okay. Uh, Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των αγορητών. Και σας ευχαριστώ. Κύριε Στομπεντίνη, παρακαλώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα σχόλια. και σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον, την συγκήτρια κυρία Καπεθών Ρουίθ, τους Ευρωβουλευτές για την συζήτηση, την ανάλυση, τους τέσσερις ομιλητές για τη δουλειά τους και το υλικό προσκέψη που μας προσέφεραν πολύ ενδιαφέροντα έννοιες, ιδέες, αριθμητικά στοιχεία τα οποία ίσως χρειάζεται να μελετήσουμε περαιτέρω. Τουλάχιστον για να καταλάβουμε καλύτερα από πού προέρχονται τα στοιχεία αυτά. Η βάση πάντως επικοινωνίας είναι πολύ καλή και ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση για την καλύτερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Δηλαδή εμεί αξιολογούμε πριν καταθέσουμε προτάσεις. Κοιτάμε προ τα πίσω λοιπόν για να προετοιμαστούμε να κοιτάμε και προ τα μπρο. Αυτή ήταν και η προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Εμείς ξέρετε κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε ένα εξελίξει μια ενδιάμεση αξιολόγηση στην οποία περιλαμβάνεται και μια φάση δημοσίων διαβουλεύσεων. Μάλιστα τώρα ε, είχα επικοινωνία με τον συνάδελφο κύριο Φαντεφνής ο οποίος μου λέει ότι έχουμε φτάσει στις 2.000 απαντήσεις στην ε, δημόσια αυτή διαβούλευση, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και δείχνει άλλωστε και την κινητοποίηση των κοινοτήτων έρευνας και κοινοτομίας. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγηση υπάρχει ένα πάνελ το οποίο θα βοηθήσει μετά την αξιολόγηση να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Είδαμε βέβαια διαφορετικές απόψεις ε, ε, που δείχνουν ότι δεν είναι στόχοι, δεν είναι αυτός η έρευνα και η καινοτομία, αλλά μέσα για την επιτεύξη στόχων. Αυτό άλλωστε ήταν και το νόημα της συζήτηση. Για να ολοκληρώνουμε, Πρόεδρε, και για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης, καταγράφουμε όλα τα μηνύματα, τα λαμβάνουμε υπόψη, λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις των μελών του πάνελ, το, το εύρος, το πλάτος, το βάθος, τον πλούτο και τη σημασία για την ε, ανταγωνιστικότητα για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ευημερία των πολιτών μας, ε, ένα σύστημα αντιμετώπισης ε, και αξιολόγησης των συνεπειών για την έρευνα και καινοτομία. Μάλιστα, λέει ευχαριστώ. Κάποιες παρατηρήσεις είχαν προσωπικό χαρακτήρα για τον κύριο Έλερ. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, αλλά παρακαλώ εν συντομία γιατί δεν έχουμε χρόνο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην, παρε... παρεξηγηθούν αυτά που υπόθηκαν, να μην, κάνουμε... να μην αντιλήσουμε λάθος συμπεράσματα. Έχουμε κάνει τη συζήτηση για το Horizon 2020 με το Γιάζι Μπούτζεκ, υποφαινόμενο συνέταξαν το πρόγραμμα συγκεκριμένα και όταν παρουσιάζουν στοιχεία που λένε ότι τα χρήματα του προγράμματος widening πάνε στα νεότερα κράτη-μέλη, που άλλωστε αυτό είναι και το νόημα του προγράμματος widening, δηλαδή είναι πρόγραμμα αδελφοποίησης, αποφασίζουν τα κράτη-μέλη αν θέλουν μια θεσμική προσέγγιση, όπως την επιλέξουν με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα Ινστιτούτο ερευνητικό, το οποίο στη συνεργασία του περιλαμβάνει την Πολωνία ή κάποιο άλλο κράτος των 13 νεότερων Βεβαίως αν πάρουμε στατιστική, στατιστικά στοιχεία μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κάποιος παίρνει λεφτά και δαπανά τα χρήματα που θα χρειαστούν για να χτίσει κάποιος άλλος ανισοτό στη χώρα του. Άρα το περισσότερα από τα στοιχεία πάνε πάλι στα 15 με την ανάλυση αυτή γιατί έχουν ε, πληρώσει αυτό που αποφάσισαν τα 13 στα προγράμματα αδελφοποίησης για την ανάπτυξη των δομών στα 13 νεότερα κράτη. Ως βάση λοιπόν κατηγοριών ότι και το πρόγραμμα Widening μπορεί να δίνει χρήματα περισσότερα στα κράτη, στα 15 παλαιότερα. Μπορεί τα στατιστικά σας να μην είναι εσφαλμένα, αλλά στην πράξη οδηγούν σε παρερμηνίες, γιατί η βασική λογική είναι ότι κάποιος πληρώνει για να χτιστεί κάτι σε ένα άλλο κράτος. Αυτό είναι το σύστημα του Widening. Εκ μέρου του ΕΛΚ λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνουμε για το widening. Εγώ θα μιλούσα ακόμη και για διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος widening, ιδιαίτερα η ομαδοποίηση, η αδελφοποίηση στοχεύει ακριβώς την ανάπτυξη των δομών στα νέα με ελληνές δομές, νέες δυνατότητες για ανταλλαγές, ώστε να απαλλαγούν από το παλαιό πανεπιστημιακό σύστημα. Και για να μην με παρεξηγείτε, αυτό που θέλω να πω απλώς είναι ότι ναι, ξέρουμε τα στοιχεία. Θα μπορούσαν να έχουν ακόμη και πιο ακραία απεικόνηση, όχι 5%, 3,9%. Είναι μειωτική η τάση και αυτό είναι θλιβερό. Αλλά με την ανάλυση, πέραν του να λέμε «Α, τα πράγματα έχουν έτσι», πρέπει να προχωράμε και να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Για μένα αν είμαστε και λίγο έντιμοι, γιατί υπήρξε μεγάλη αντίσταση από τα 13 νεότερα και όχι όλα βέβαια, ε, κράτη-μέλη, μεγάλη αντίσταση στην επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία, γιατί έλεγαν Θέλουμε τα χρήματα για τα διευθυντικά ταμεία, το έλεγαν στο Συμβούλιο και μέσα από τα διευθυντικά ταμεία η Επιτροπή μας, μαζί με την Επιτροπή της Ιστορικής Αγοράς, ψήφισε για να παραμείνει η έρευνα και η τεχνολογία κατά ένα τρίτο στο διευθυντικό ταμείο. Και αν δείτε τον κατάλογο των ψηφοφοριών του Συμβουλίου και των δικών μας, θα αντιληφθείτε ότι τα 15 παλαιότερα κράτη-μέλη και η τελευταία ε, πολωνική κυβέρνηση υπερψήφισαν την πρόταση αυτή και όλα τα άλλα από τα νεότερα κράτη-μέλη ψήφισαν. Τώρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Η ανάλυση για οποιαδήποτε πίεση θα μπορούσε να εκφραστεί και τάσεις για το πρόγραμμα πλαίσιο 9. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θέλουν περισσότερη συμμετοχή. Αν όμως συνεχίσετε με αυτές τις ε, ε, ε κατηγορίες, δεν μπορώ να βρω λύση γιατί και το Συμβούλιο με τα νεότερα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο μιλούν μόνο για μισθούς, τίποτε περισσότερο. Πρέπει λοιπόν από κοινού να αναζητήσουμε μια λύση και να μην περιπέσουμε στην επανάληψη τετριμένων κατηγοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τον κύριο καθηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μεγάλος κατάλογος ερωτήσεων και βεβαίως ίσως να μην καταφέρω να τις απαντήσω όλες, αλλά κάποιες παρατηρήσεις για ορισμένα ζητήματα πρέπει οπωσδήποτε να τα ε, θίξουμε. Καταρχάς είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια Καμπεθών Ρουίχ που τόνισε τη σημασία της συμμετοχής ε, Τα προγράμματα όπως το πρόγραμμα πλαίσιο δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ε, αριστεία, αλλά θέλω να εξασφαλίσουν ότι αυτή οι θύλακη αριστείας σε διάφορα σημεία τη Επιπύρου εντοπίζονται. Ο κόσμος να ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε διάφορε ερευνητικέ ομάδε και ιδρύματα ε, που μπορούν επίση να συμμετέχουν και αυτό είναι τρόπο να ε, ξεπεραστεί και το θέμα τη ανισότητα. Να μιλάμε για την αριστεία που είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι έχουμε πολλέ ωρε σκημωμένες σε διάφορες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Όταν δει κανείς τη στατιστική, τις για το ορίζοντας 2020 δεν το πιστεύει ότι υπάρχουν αυτές, ε, αλλά υπάρχουν. Κάποιοι δεν θέλουν απλώς να το ανακαλύψουν. Μπορεί να βρουν μια πριγκίπισσα ε, όπου ο ο ωραίος πρίγκιπας θα τις ερωτευτεί. Πάντως το πρόβλημα είναι ότι για, τη για την ώρα είναι κλεισμένοι σε, οι, πριγκίπι, πριγκίπισσες αυτές είναι κλεισμένες σε πύργους και κανείς δεν θέλει να τις συναντήσει. Uh, Mr. Eller was, uh, was kind enough to mention that uh, members of European Parliament are waiting. Οι Ευρωβουλευτές ε, περιμένουν συγκεκριμένες προτάσεις ε, και θα σας τονίζω τρία σημεία που αφορούν ε, τρόπους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά και το, τη λογική Γιατί όταν υποβάλλονται οι προτάσεις ακούμε ότι πρόκειται για την ίδια συζήτηση, ότι δηλαδή ξαναπέφτουμε σε θέσεις που εκφράστηκαν πριν από πέντε χρόνια. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα σχεδιασμού του στο ορίζοντας 2020, ε, ε, ότι δηλαδή δεν προέβλεψε την ενεργή συμμετοχή ορισμένων ομάδων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, ε, πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξηθεί η συμμετοχή, αλλά αντίθετα για την ώρα γίνεται όλο και χειρότερη κατάσταση. Με τα, στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε, τα επίπεδα συμμετοχής μειώνονται για τις 13 χώρες. Γιατί να μην αρχίσουμε να εξετάζουμε λοιπόν τα στοιχεία, να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε τη συζήτηση για κάποιον ιδεών, αντί να λέμε ότι πριν από πέντε χρόνια σκεφτόμασταν κάτι και τώρα δεν θέλουμε να αναθεωρήσουμε τις ε, Εγώ θέλω να σας παροτρύνω να δείτε προσεκτικά τα στοιχεία και να σκεφτείτε πως ίσως υπάρχει τρόπος να αναθεωρήσουμε κάποια στοιχεία σχεδιασμού του προγράμματος. Επιπλέον ανάλυση λοιπόν. Η κυρία Σκιώδης εισηγητή Κουντρίτσκα ανέφερε ότι η διάδοση και η επέκταση της συμμετοχής είναι μεγάλη πρόκληση. εννοώ να συμφωνήσω γιατί είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχουν ε, ε, αδελφοποιήσεις ε, έχουμε τέρους από διαφορετικές χώρες αλλά ταυτόχρονα μήπως θα πρέπει να διευρυνθεί και το πακέτο των κέντρων αριστείας ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν και τα κέντρα αριστείας ε, των, της, του, ε13 γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία. 52% 52% του προπολογισμού πάει στις χώρες της EU15. Ε, είναι πρόβλημα. Logic of of a twinning program is that you pay Η λογική είναι ότι πληρώνεις για ένα Ινστιτούτο που πρέπει να οικοδομηθεί στη χώρα σας. Αυτό δεν είναι παράδειγμα για το ότι πάντα χρήματα στην, στην, στην Ένωση των 15. Όχι, θέλετε να, πολύ περισσότερα. Μα με αυτό δεν το έχουμε όμως συμφωνήσει. Η λογική, τα νούμερα, πώς μπορείτε να λέτε ότι η διεύρυνση είναι ένα, τρόπο, ένα, ένα, ένα παράδειγμα ε, για το ότι τα χρήματα της διεύρυνσης πάνε στην ε, ε, Ένωση των 15. Κοιτάξτε, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, ε, μετά τη συνεδρίαση, γιατί ίσως θέλει πιο ισότερη συζήτηση αυτό. Μάλιστα, να, πιο σύντομα. Κύριε Σκιώδη, ο, ο μάλλον ο Σκιώδης, ο κύριος Μαραγκάλα ανέφερε ότι εντός ομάδων χωρών μέσα ε, στην Ένωση των 15 ή των 13 έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις χωρών ή περιφερειών που μπορεί να μείνουν απ' έξω για ορισμένα δίκτυα και προγράμματα. Συμφωνώ και αυτό είναι θέμα που μάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί όταν μιλάμε για τον σχεδιασμό του ένα του προγράμματος πλαισίου. Η κυρία Βιέρνιγκ αναφέρεται την ανησυχία της για την ε, χρηματοδότηση της δικτύωσης στο Horizon 2020. Ίσως να χρειαστεί να εξηγήσουμε και πάλι τη δήλωση Πρέπει να ανοίξουν τα δίκτυα, όχι μόνο να δώσουμε χρηματοδότηση χρηματοδότηση για μετακίνηση για την παρακολούθηση συνεδριάσεων, ίσως να μην είναι αυτό το θέμα. Το πιο σημαντικό είναι όταν υπάρχει εξαιρετική έρευνα, αλλά Κάποιοι εταίροι των ε, συμπράξεων μπορεί να προτιμούν να παραμείνουν και να συνεργαστούν με τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκαν για πολλά χρόνια. Οπότε, αν ε, στραφούμε στο θέμα που, μάλλον το σχόλιο που διατυπώθηκε από την κυρία Νίμπλερ, που δεν είναι πια στην αίθουσα, αν έχουμε θετικά παραδείγματα επιτυχίας για το Horizon 2020 και τα προγραμματά του από τις χώρες ε, το 13, ναι, η έρευνα ε, στο δικό μου πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Βασοβίας είναι ο πρώτος δικαιούχος ε, φορέας της Πολωνίας και μπορώ να σας πω ε, στα ίσια ότι έχουμε μεγάλα εμπορι... μεγάλες εμπορικές και καινοτόμες επιτυχίες projects τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Εθνική Χρηματοδότηση, από τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης και δεν έχουμε ούτε μία περίπτωση που χρηματοδόθηκε από το, από το πλαίσιο 8, 7 από το ορίζον 2020. Ε, ίσως αυτό να σχετίζεται με το γεγονός ότι είχαμε πιο εύκολη πρόσβαση σε μεγάλους προπολογισμούς έρευνα και ανάπτυξη που μοιράστηκαν στους, στους που ήταν επιτυχείς και που αποκρίνονταν στα διεθνή κριτήρια σύγκριση ομοτήμων. Μάλιστα. Είναι σημαντικό, κύριε καθηγητά, να λάβετε υπόψη ότι για τα κράτη-μέλη έχουμε πάνω από 90% χρηματοδότηση για την έρευνα. Το πρόγραμμα πλαίσιο 7 είναι λιγότερο από το 10%. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη είναι πάντοτε το ίδιο. Ένα είναι το πρόγραμμα πλαίσιο και νέα είναι ε, το ίδιο το κράτος. Αυτό θα πρέπει να το θυμηθούμε. Ο κύριος Σαν Σεμπαστιάν. Ευχαριστώ. Δεν υπήρχαν και πολλά ερωτήματα για μένα από ό,τι φαίνεται. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, αλλά θυμάμαι πριν από 30 χρόνια περίπου όταν η Ισπανία άρχισε να συμμετέχει στο πέμπτο πρόγραμμα τότε και εμεί είχαμε ένα θέμα το πώς θα συμμετάσχουμε ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Και κάναμε ένα άλμα τότε. Μάθαμε. Υπήρξε μια διαδικασία εκμάθησης με την υποστήριξη των περιφερειακών κυβερνήσεων της εθνικής κυβέρνησής μας που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και, στην ένατη, και στο ένατο πλαίσιο. Θα πρέπει να επιταχυνθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία. Βεβαίως ε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας δώσει συμβουλές για το πώς θα το καταφέρετε αυτό. Πάντως ε, έχουμε πολλές επιτυχείς συνεργασίες με ερευνητές από τις χώρες αυτές, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Κάποια από αυτά που είπα μάλλον παρεξηγήθηκαν, παρανοήθηκαν και να το εξηγήσω. Βεβαίως και η βασική έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική εάν θέλουμε να είμαστε μια καινοτόμος περιοχή του κόσμου. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλησα να πω κάτι άλλο. Εγώ είπα ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα διάφορα στάδια της έρευνας. Από τη βασική έρευνα έως την αγορά. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα κλειδί. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι μοχλοί όθησης στο καθένα από αυτά τα στάδια θα πρέπει να δούμε πού βρίσκονται τα κενά, πού η διαδικασία αυτή δεν λειτουργεί. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε κατά νου το σύνολο της διαδικασίας. Το ερώτημα για τον αντίκτυπο τώρα. Εφόσον μιλάμε για τα τεχνολογικά κέντρα, τα RTOs, ε, το κάθε RTO έχει το δικό της πεδίο επιρροής, δικό του πεδίο επιρροής. Και βεβαίως ε, άλλα είναι ευρύτερα, άλλα πιο περιορισμένα, άλλα είναι εθνικά, άλλα περιφερειακά, αλλά εξαρτάται πάντα από το πεδίο ε, στο οποίο εργάζονται και στην περιοχή στην οποία εργάζονται ο αντίκτυπος. Οι περιοχές εκείνες όπου υπάρχουν ισορροπημένα οικοσυστήματα, εκεί είναι που συμβαίνουν πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας αυτήν την ιδέα του να φτιαχτούν οικοσυστήματα, το να, έχει, να έχουμε δηλαδή ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Δεν είναι επαρκές. Ούτε το να υπάρχουν κεφάλαια είναι επαρκές, ε, κεφάλαια κινδύνου. Όχι, χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται ένα οικοσύστημα ισορροπημένο, ε, συνδεδεμένο με άλλα. Για το ερώτημα του κατά πόσο θα άλλαζα το σύστημα αξιολόγησης. Ναι, θα το άλλαζα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος όλων των προτάσεων αυτών, όλη αυτή τη διαδικασία υποβολή προτάσεων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελαχιστοποιήσουμε το έργο που επιτελούμε για να φτάσουμε σε αυτέ τι καλέ προτάσει. Χρειάζεται μια αξιολόγηση σε δύο στάδια και αφού γίνει όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, να βρεθούν μέσα για να εκμεταλλευτούμε αυτό το έργο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την εκπληκτική αυτή συζήτηση. Όλοι σας, αναλυτές, ομιλητές, ε, υποβάλλατε προτάσεις ε, έντονες. Ε, μιλήσαμε για το ένα το πρόγραμμα. Από την άλλη, οι συνάδελφοι από το Ευρώπινο Βούλιο συμμετείχαν και αυτοί. Πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διότι αισθανόμαστε υπεύθυνοι για το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο, όχι για την διάμεση αξιολόγηση του ορίζοντα 2020. Σας ευχαριστώ πολύ για την καταπληκτική συζήτηση και για τον χρόνο που αφιερώσατε σε, σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής. Φέτος, κάθε φορά συζητούσαμε το θέμα αυτό. 12 Ιανουαρίου η επόμενη συνάντηση, 9 το πρωί, για 3,5 ώρες. Τελευταία συνάντηση, τελευταία συνεδρίαση πριν το τέλος της ε, μισής θητείας μας. Μισή θητεία, έτσι. Απίστευτα το πώς πέρασε ο καιρός. Είναι απογοητευτικό για μένα αυτό, αλλά είναι καλό νέο. Υπάρχει ένα καλό νέο για όλους, ότι έχουν τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Λοιπόν, θα, νομίζω θα πιούμε και ένα ποτό χριστουγεννιάτικο. Οπότε δεν σα λέω, δεν λέω χρόνια πολλά, δεν σας λέω καλά Χριστούγεννα ακόμα, μόνο στους ε, προσεγγλημένου εδώ. Λοιπόν, 12 Ιανουαρίου η επόμενη συνάντηση και βεβαίως μην ξεχνάμε και το χριστουγεννιάτικο ποτό που θα πιούμε. Ευχαριστώ.